Αγαπητοί συνάδελφοι, είναι 9 και 7 και 8. Ας αρχίσουμε, ακόμη και αν τα νέα της ημέρας μας κινούν και πρέπει να σκεφτούμε φυσικά πως τα αποτελέσματα των εκλογών στις Ηνωμένες Πολιτείες θα έχουν επιπτώσεις στο παγκόσμιο σύστημα εμπορίου και στις δικές μας σχέσεις με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό σίγουρα θα αποτελέσει θέμα συζήτησης σε μία από τις επόμενες συνεδριάσεις, ίσως και στην επόμενη. Κατά την άποψή μου, οι εκλογές αυτές σημαίνουν μία θεμελιώδη αλλαγή πορεία στην εμπορική πολιτική των ΗΠΑ αν ένα μέρος μόνο των εξαγγελιών του κυρίου Τραμπ υλοποιηθεί, δηλαδή αν έχουμε απομονωτισμό και εμπορικό πόλεμο με την Κίνα. Όλα αυτά θα αλλάξουν το παγκόσμιο κλίμα σαφώς και πρέπει να στοχαστούμε πολύ γρήγορα για την στάση την οποία θα έχουμε απέναντι στο θέμα αυτό. Παρά τα αυτά έχουμε την ημερήσια διάταξη όπως την έχετε λάβει. Έχω τρεις προτάσεις τροποποίησης. Και μάλιστα υπάρχει η ψηφοφορία για την μακροοικονομική στήριξη της Ιορδανίας το σημείο 15, αυτό μπορούμε να το μεταθέσουμε μετά το 21. Υπάρχει η πρόταση της κυρίας Μόσκα, της εισηγήτριας, να εισαχθεί μια προφορική ερώτηση την οποία θα εισάγουμε στις ψηφοφορίες και σχετικά με την έκθεση για την επίσκεψη στη Βαλένσια, σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης, μπορεί επίσης να μετατεθεί πιο σε ένα αργότερο χρονικό σημείο. Υπάρχουν ενστάσεις, αντιρρήσεις ενάντια στις αλλαγές αυτές ή στην ημερήσια διάταξη. Όχι, δεν έχουμε, οπότε εγκρίνεται η ημερήσια διάταξη. Σημείο 2, έγκριση των πρακτικών και εδώ θα προχωρήσουμε ως εξής. Αν δεν υπάρξουν αντιρρήσεις για τα πρακτικά έως το τέλος της συνεδρίασης, τότε τα πρακτικά θα εγκριθούν ως έχουν. Σημείο 3. Ανακοινώσεις του Προέδρου. Πρώτα απ' όλα υποδεικνύω πάντα στην αρχή πως και αυτή η συνεδρίαση μεταδίδεται ζωντανά μέσω ίντερνετ, οπότε χαιρετίζω ήδη όλους τους τηλεθεατές μας από τη Λιουμπλιάνα έως το Ελσίνκι και τις άλλες ευρωπαϊκές πόλεις. Χαίρομαι πολύ που έχουμε τόσους τηλεθεατές μέσω διαδικτύου, αλλά μην ξεχνάτε αναμεταδίδεστε διαρκώς. Κάποιες ανακοινώσεις ακόμα. γνωρίζετε πως η θητεία του Γενικού Γραμματέα του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, του κυρίου Αζεβέντο, λύγει το 2017. Ο κύριος Αζεβέδο δήλωσε ωστόσο πως θα υποβάλει εκ νέου υποψηφιότητα ως Γενικός Γραμματέας. Αυτό είναι θεωρητικά δυνατόν και πρακτικά. Ο Πασκάλ Λαμίν είχε επίσης δύο θητείες Εάν υπάρξουν νέοι υποψήφοι, αυτοί πρέπει να υποβάλουν την υποψηφιότητά τους μεταξύ 1ης και 31ης Δεκεμβρίου και στη συνέχεια οι υποψηφοί έχουν τρεις μήνες καιρό για να συστηθούν και η οριστική απόφαση θα ληφθεί την 31η Μαΐου 2017. Έως τώρα δεν άκουσα για κάποιους άλλους υποψηφίους, αλλά κανείς δεν ξέρει. Επίσης υποδεικνύω πως είχαμε μια πολύ επιτυχή αποστολή στη Αργεντινή. Θα το συζητήσουμε σύντομα σε ένα ξεχωριστό σημείο της ημερήσιας διάταξης και όλοι μας γνωρίζουμε πως του χρόνου τον Μάιο είναι οι προεδρικές εκλογές στη Γαλλία και σε ένα μικρότερο κόμμα, στους πράσινους, ένας συνάδελφος από αυτή την επιτροπή, ο Τζανίκ Τσαντό, είναι υποψήφιος πρόεδρος της Δημοκρατίας εκ μέρους των Πρασίνων. Ήθελα να σας το ανακοινώσω στο πλαίσιο μιας δίκαιης αντιπαράθεσης και αυτού που θεωρώ πολιτικά δίκαιο. Εύχομαι σε προσωπικό επίπεδο καλή επιτυχία. Πολύ ωραία. Οπότε περνούμε στο σημείο 4. Επί του παρόντος έχουμε δύο τριμερείς διαλόγους. Ο ένας πραγματοποιείται σε σχέση με την ολοκλήρηση της νομοθεσίας σχετικά με τα ορυκτά συγκρούσεων. Βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ελπίζω να μπορέσουμε να το ολοκληρώσουμε στο εγγύς μέλλον. Πρέπει να αποσαφηνίσουμε κάποια τεχνικά ζητήματα. Ο εισηγητής μου κάνει νόημα πως βρισκόμαστε όντω σε πολύ καλό δρόμο. Ορίστε. Ποιες συγκρούσεις υπάρχουν ακόμα ή έχουν επιληθεί όλα τα ουσιώδη ζητήματα. Κάποιες λεπτομέρειες ακόμα. Τα ουσιώδη ζητήματα έχουν επιληθεί. Το ζητούμενο είναι τώρα μόνο πως προβήκαμε στην παραχώρηση πως για μικρούς εισαγωγείς θα υπάρξουν εξαιρέσεις. Απλά η, η ταυτοποίηση αυτού, δηλαδή τι σημαίνει αυτό ακριβώς, για ποια ποσοστά μιλάμε, για ποιους όγκους, αυτό, είναι, αυτό μας απομένει να αποσαφηνίσουμε. Όλα τα άλλα ερωτήματα, όπως τα κριτήρια, οι κατευθυντήριες γραμμές, για αυτά έχουμε επιτύχει συμφωνία. Ευχαριστώ Μπέρντ. Είναι πολύ σημαντικό που υποδεικνύουμε πως με την ομοθεσία πηγαίνουμε ένα βήμα προς τα μπροστά υπό την έννοια της επιχειρηματικής ευθύνης και πως καθιστούμε σαφές πως η εμπορική πολιτική μπορεί να συνεισφέρει στην επίλυση συγκρούσεων. Χθες το βράδυ υπήρξε μια ταινία στη γερμανική τηλεόραση στην οποία έλαβε το λόγο εσύ επίσης στην οποία παρουσιάστηκε ο κανονισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκεί έγινε σαφές πως κάνουμε ένα πρώτο βήμα και πως εμείς ως Κοινοβούλιο θα πρέπει να συνεχίσουμε να εργαζόμαστε στην μεταξέλιξη της νομοθεσίας αυτής. Πρέπει δηλαδή να διασφαλίσουμε αυτό που επιτύχαμε, επίσης κατά της αντίστασης κάποιων κρατών μαλλιών και πρέπει να ασκήσουμε πίεση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ο εισηγητής μας Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. Υποστηρίζω πλήρως αυτά που είπατε βεβαίως και το γεγονός ότι τα προβλήματα τα οποία ακόμα πρέπει να επιλύσουμε δεν είναι τα σοβαρά προβλήματα. Υπάρχουν κάποιες ε, λεπτομέρειες ίσονος σημασίας, σημαντικές ένα, αλλά ακόμα λεπτομέρειες, για τις οποίες ε, βεβαίως νομίζω ότι ε, βρισκόμαστε στην καλύτερη δυνατή θέση για να τι επιλύσουμε. Θα ήθελα λοιπόν να επαναλάβω τη δήλωσή σα. Η αίσθηση δική μου ως εισηγητή είναι ότι κατά πάσα πιθανότητα στις 22 Νοεμβρίου στο Στρασβούργο θα μπορέσουμε να έχουμε τον τελευταίο τριμερή διάλογο, ο οποίο θα οριστικοποιήσει τα πράγματα, αν όλα πάνε καλά βεβαίω. Θα γίνει μια πρώτη εσωτερική συνεδρίαση για να συντονίσουμε τα τελευταία των διαπραγματεύσεων το πρωί με την διαπραγματευτική ομάδα και τις πολιτικές ομάδες και αυτό το οποίο θα ήθελα να επισημάνω είναι ότι η πολιτική συνεννόηση στην οποία καταλήξαμε το καλοκαίρι έχει γίνει πλήρως σεβαστή. Επομένως προχωρούμε και στις κατευθυντήριες γραμμές και βάση της πολιτικής συνεννόησης και ε, θα ήθελα να αποτίσω φόρο τιμής για άλλη μια φορά στην Ολλανδική Προεδρία, διότι ο εταίρος του Κοινοβουλίου στον τριμερή διάλογο αυτό το καλοκαίρι ήταν η Ολλανδική Προεδρία και πρέπει να του συγχαρώ για τη δραστηριότητά τους και ε, θα ήθελα να το κάνω και ε, για τη Σλοβακική Προεδρία, διότι πιστεύω ότι αν υπάρξει η ίδια αποφασιστικότητα, τότε σίγουρα στις 22 Σεπτεμβρίου θα μπορέσουν να οριστικοποιήσουμε το ζήτημα και αυτό ε, σημαίνει ότι θα γίνει και εντός της Σλοβακικής Προεδρίας, επομένως θα έχουμε ένα καλό αποτέλεσμα. Ευχαριστώ. Äh, ευχαριστώ πολύ κύριε Βίνκλερ, σας ευχαριστώ επίσης όλους σας επειδή γνωρίζουμε πως στην αρχή είχαμε διαφωνίες εδώ στο Κοινοβούλιο, αλλά τώρα ως διαπραγματευτική ομάδα έχουμε επιτύχει μια συνοχή και παρουσιαστήκαμε με μια φωνή και πιστεύω πως αυτό είναι μια μεγάλη επιτυχία. Και αυτό που είπε και ο κύριος Σόλτς είναι πως το νομοθετικό πακέτο που έχουμε τώρα είναι κάτι εντελώς καινούριο και πως αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για μια δίκαιη διαμόρφωση του εμπορίου με πρώτες ύλες. Έτσι στις 22 Νοεμβρίου στο Κοινοβούλιο, στην ολοκλήρωση της διαδικασίας, μπορούμε να είμαστε πολύ περήφανοι για τις επιδόσεις μας, οι οποίες είναι σημαντικές. Δεύτερος τριλόγος. Η μακροοικονομική στήριξη της Ιορδανίας γνωρίζετε, το αποφασίσαμε πρόσφατα στην Επιτροπή. Υποστηρίζουμε καταρχάς την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Αυξήσαμε το ποσό από τα 200 εκατομμύρια στα 350 και προβήκαμε σε κάποιες τεχνικές τροποποιήσεις τις οποίες προτείναμε. Στις 27 Οκτωβρίου είχαμε έναν τριμερή διάλογο στον οποίο κατέστη σχετικά γρήγορα σαφές πως το Συμβούλιο σε καμία περίπτωση δεν θέλει να αυξήσει το ποσό των 200 εκατομμυρίων. Οπότε κατά βάση για τη διαπραγματευτική μας ομάδα είχαμε την επιλογή είτε να διακόψουμε τον τριμερή διάλογο χωρίς προοπτική να υπάρξει κάποια κίνηση από την πλευρά του Συμβουλίου εν ώψη της δημοσιονομικής κατάστασης ή να, ή να επιδιώξουμε μια κοινή δήλωση του Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής με μια σαφή δήλωση πως εάν τα, ε, εφόσον είναι δυνατόν να λάβει η Ιορδανία την μακροοικονομική στήριξη. Πρόκειται για μια πολύ ξεκαθαρή διατύπωση την οποία επιδιώξαμε πολύ στεναρά. Αυτή ήταν η επιλογή την οποία μπορούσαμε να επιτύχουμε και επίσης διασφαλίσαμε αυτή η κοινή δήλωση μαζί με το νομοθετικό πακέτο να δημοσιευτεί στην επίσημη εφημερίδα. Πιστεύω πως και τα δύο είναι μια αποδεκτή επιτυχία. Αφενός, τώρα η υποστήριξη μπορεί, η στήριξη αυτή μπορεί να υλοποιηθεί και αφετέρου έχουμε την επιλογή πως εάν χρειαστούν περισσότερα χρήματα αυτά μπορούν να παρασκεθούν. Γι' αυτό και μπορούμε να προβούμε σε μια ψηφοφορία επί του συμβιβασμού. Ωραία. Οπότε περνάμε στο πέμπτο σημείο. Είναι η έκθεσή μας από την αντιπροσωπεία στο Buenos Aires και για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης χαιρετίζω επίσης εκπροσώπους της Αργεντινής Πρεσβείας που βρίσκεστε. Α, μάλιστα. Καλώς ήρθατε. Ορίσαμε την αντιπροσωπεία και πραγματοποιήσαμε την αποστολή της επειδή ήμασταν πεπισμένοι πως μετά από την ανταλλαγή προσφορών στις 11 Μαΐου για τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Μερκοσούρ και Ευρωπαϊκής Ένωσης τον πρώτο πραγματικό κύκλο διαπραγματεύσεων από το 2012, τον Οκτώβριο του 2016, οι επιλογές για μια ενισχυμένη διαπραγματευτική διαδικασία πληρούνται και πως ήμασταν επίσης της άποψης πως υπό το πρίσμα της αθεροποίησης του κυβερνητικού έργου στην Αργεντινή μπορούμε, θα έπρεπε να αποστείλουμε μια τέτοια αντιπροσωπεία το οποίο και κάναμε. Και όπως πάντα η αντιπροσωπεία μας αφενός ήταν πάρα πολύ καλά προετοιμασμένη, ευχαριστώ πάρα πολύ την γραμματεία γι' αυτό. Όλες οι συναντήσεις, όλη η επιμελητεία, όλα λειτουργήσαν πολύ καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ γι' αυτό. Αλλά είχαμε επίσης τη δυνατότητα να συζητήσουμε με υπεύθυνου πολιτικούς συχνά σε πολύ υψηλό επίπεδο. Μεταξύ άλλων συναντηθήκαμε με την Υπουργό Εξωτερικών κυρία Λόρκα, τον Υπουργό Οικονομίας επί μία ώρα πολύ έντονα για οικονομικά ζητήματα με τον Υπουργό Εργασίας και τον Υφυπουργό Εμπορικών Ζητημάτων με τον οποίο είχα τη δυνατότητα να συζητήσω και εδώ στις Βρυξέλλες. Επρόκειτο για έναν πολύ επικοδομητικό και ευχάριστο διάλογο, αλλά επίσης συναντηθήκαμε με εκπροσώπους του Κοινοβουλίου, της κοινωνίας των πολιτών, δεξαμενών σκέψης, εκπροσώπους του αγροτικού τομέα, επειδή πιστεύω πως ο αγροτικός τομέας αποτελέσει σημείο κεντρικής σημασίας κατά τις διαπραγματεύσεις. Έτσι αποκτήσαμε μια εκτενή εικόνα για το πώς η Αργεντινή μπορεί να διαμορφώσει τις διαπραγματεύσεις με την Μερκοσούρ αλλά και πώς οι διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να συνεχιστούν προς το συμφέρον μιας εκτενούς συμφωνίας και είμαι πεπισμένος πως υπό το πρίσμα της κατάστασης που είδαμε σήμερα στις Ηνωμένες Πολιτείες, τέτοιες συμφωνίες είναι πολύ σημαντικές για να καθορίσουμε κανόνες. Κατά την απόψή μου, δηλαδή μια πολύ επιτυχής αντιπροσωπεία, κάποια από τα μέλη της βρίσκονται εδώ μαζί μας, ο εισηγητής κ. Σάλμπα. Θέλετε να συμπληρώσετε κάτι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Το είπατε κι εσείς ε, πριν από δύο μέρες επιστρέψαμε από την επίσημη αποστολή της Επιτροπής μας στην Αργεντινή. Νομίζω ότι όλοι εκείνοι που συμμετείχαν μπορούν να θεωρήσουν ότι ήταν πολύ ε, παραγωγική και αποτελεσματική. Η αντιπροσωπεία θα υποβάλει και γραπτή έκθεση εντό του μηνό, αλλά πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό, το είπε και ο Πρόεδρο, να εκμεταλλευτούμε αυτή την ευκαιρία και να πούμε στου συναδέλφου ε, την άποψή μα και την εικόνα που αποκομίσαμε ε, στη διάρκεια αυτή τη αποστολή. Το είπε ο Πρόεδρο, πρόκειται για μια αποστολή ε, αρκετά πυκνή, διότι σε δυόμιση μέρε ε, συναντηθήκαμε με έναν κατάλογο συνομιλητών ε, πολύ υψηλού επίπεδου που μας περιέγραψαν ε, την κατάσταση στην Αργεντινή, τις προκλήσεις, ε, τις ευκαιρίες που προσφέρει η χώρα και ε, τα στοιχεία τα οποία θεωρούν ότι είναι τα πιο σημαντικά στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ. Όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, συνεδριάσαμε με υπουργούς, τεχνικούς, συνομιλητές, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, και είχαμε πολύ συγκεκριμένε ε, συνεδριάσεις ε, με την κοινότητα της υπαίθρου της Αργεντινής, ε, συνομοσπονδίες σωματείων της Αργεντινής και είναι αλήθεια ότι υπήρξε μεγάλος ενθουσιασμός και αισιοδοξία όσον αφορά την επίτευξη αυτής της συμφωνίας και επίσης να πω ότι το βιομηχανικό επιμελητήριο της ε, Αργεντινής ήταν λίγο πιο επιφυλακτικό όσον αφορά τις δυνατότητες της, ε, ε, της βιομηχανίας της Αργεντινής να ανταγωνιστεί την ευρωπαϊκή βιομηχανία αυτή τη στιγμή υπογραφή συμφωνία. Κάναμε και κάποιες τεχνικές συνεδριάσεις για την ε, εξέλιξη των εμπορικών ε, ε, σχέσεων και κάναμε και κάποιες επισκέψεις επιτόπου για να δούμε πώς λειτουργούν ευρωπαϊκές επιχειρήσεις οι οποίες εδρεύουν στη χώρα. Σε γενικές γραμμές θεωρώ ότι όλοι οι συνομολητές μας, αλλά και εμείς, αντιλαμβανόμαστε ότι πρόκειται για ιστορική στιγμή και ε, ότι υπάρχει ανάγκη να υπάρξει μια κοινή στρατηγική η οποία θα ενισχύσει τις ανταλλαγές απόψεών μας σε όλους τους τομείς. Η ενίσχυση του εμπορίου και η ε, ανάπτυξη των επενδύσεων είναι κάτι το οποίο όλοι θεωρούν ε, ομόφωνα ότι θα επιτευχθεί. Πρόκειται για ιστορική στιγμή και νομίζω ότι έτσι προσεγγίζουμε περισσότερο και την πλευρά της Μερκοσούρ για τις επικείμενες διαπραγματεύσεις και ίσως ε, και ε, να θεωρήσουμε ότι είναι πιθανό να επιτευχθεί αυτή η πολύ σημαντική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μερκοσούρ. Δεν έχω καμία αμφιβολία ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολλά να κερδίσει από αυτή τη συμφωνία. Και ε, η πλευρά του Μερκοσούρ βεβαίως, αλλά εμείς πρέπει να κάνουμε αξιολόγηση από την ευρωπαϊκή οπτική. Θεωρώ ότι το γεγονός ότι οι οικονομίες μας αλληλοσυμπληρώνονται και ότι ο παραγωγικός μας ιστός αλληλοσυμπληρώνεται και υπάρχει και κάτι πολύ σημαντικό. Έχουμε κοινέ αξίες οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές και για το Μερκοσούρ αλλά και για την Αργεντινή πιο συγκεκριμένα και επομένω μπορούμε να θεωρήσουμε ότι είναι εταίροι ε, πάρα πολύ σημαντικοί για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύω ότι οι διατλαντικοί δεσμοί, ε, διότι όπως είπε και ο Πρόεδρος, ε, οι σχέσεις αυτές αμφισβητούν περισσότερο ε, από ποτέ μετά τα σημερινά αποτελέσματα και θεωρώ ότι οι σχέσεις αυτές δεν είναι τυχαίες ούτε συγκυριακές. Είναι καρπός μιας σύμπτωσης σε πάρα πολλούς τομείς. Κοινέ αξίες, συνήθειες και σε κάποιες χώρες ακόμα και κοινή γλώσσα τα μέλη της Επιτροπής που συμμετείχαν στην αποστολή αντιμετώπισαν ανοιχτές πόρτες για διάλογο στα Υπουργεία, στην Προεδρία, στο Υπουργείο Εξωτερικών Υποθέσεων, Οικονομικών, Οικονομίας, ε, Απασχόλησης, Γεωργίας κλπ. που επισκεφθήκαμε. Επίσης, ε, είδαμε τι προσπάθειες κάνει η κυβέρνηση του Πρόεδρου Μάκρη που ε, βρίσκεται εδώ και ένα χρόνο περίπου πλέον στην κυβέρνηση, προσπαθεί να περάσει διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ώστε να προωθήσει ε, την οικονομική βιώσιμη ανάπτυξη στην Αργεντινή και να μπορέσει έτσι να ε, βελτιώσει και τις σχέσεις του και να έχει επενδύσεις και εμπορικούς εταίρους και να βελτιώσει και την ανταγωνιστικότητα της χώρας που είναι πάρα πολύ απαραίτητη για να μπορέσει να ανταγωνίζεται επίσης όρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πιστεύουμε ότι δεν θα είναι εύκολο, διότι η χώρα την τελευταία δεκαετία είχε έναν ιδιαίτερο τρόπο να αντιμετωπίζει το εξωτερικό εμπόριο, το οποίο όπως οι περισσότεροι συνάδελφοι γνωρίζουν οδήγησε σε ε, προσκόμματα σε εμπορικό επίπεδο και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή ακόμα και η αντιπολίτευση ε, και η κοινωνία των πολιτών ε, έχουν ένα πνεύμα επικοδομητικής κριτικής και ελπίζουμε ότι αυτό θα επιτρέψει στην κυβέρνηση Μάκρη να κάνει τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις αυτή η ανάγκη πολιτικής υποστήριξης προς την κυβέρνηση Μάκρη διαβιβάστηκε και προς την ε, αποστολή μας. Μας ζήτησαν και χειρονομίες, όχι μόνο να ε, πούμε ότι υποστηρίζουμε την κυβέρνηση και τη θετική της τάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι πολύ πιο θετική από ό,τι στο παρελθόν, και μας ζήτησαν και πράξεις, επαναλαμβάνω, όχι μόνο ε, θεωρητική υποστήριξη και νομίζω ότι υπήρχε σχεδόν ομόφωνη, ομόφωνη υποστήριξη από πλευράς κυβέρνησης και εγώ προσωπικώς και νομίζω και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι θεωρούν ότι είναι ε, λογικό ε, διότι θέλουν να εφαρμόσουν το συντομότερο δυνατόν τις αποφάσεις ε, που επηρέασαν πάρα πολύ την Αργεντινή για τα θέματα αυτά. Θεωρώ ότι και η δική μας στάση θα αποτελέσει μια πολύ σημαντική χειρονομία από πλευράς ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων, να δείξουμε δηλαδή ότι υποστηρίζουμε μια κυβέρνηση που κάνει πολύ μεγάλη προσπάθεια και επομένως μέσα σε αυτό το πλαίσιο προσπάθησε να συσφίξει και τις σχέσεις ε, με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πρόκειται για τον πιο ευρωπαϊστή, αν θέλετε, ε, πρόεδρο της Αργεντινής σε σχέση με τους προηγούμενους και πρέπει να δείξουμε και εμείς την πολιτική μας υποστήριξη, ώστε η επιθυμία τους να προσεγγίσει η Αργεντινή και το Μερκοσούρ εν γέννη την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, να μην αποδειχθεί λανθασμένη και να μην απογοητευτεί ο λαός. Επίσης, συναντηθήκαμε και με σημαντικούς εταίρους και θεωρώ ότι πρέπει να υποστηρίξουμε όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ε, επρόκειται για μια ε, παραγωγική και επικοδομητική αποστολή κατά την άποψή μου και πιστεύω ότι θα δείξει ότι ε, θα μπορέσουμε στη συνέχεια να αναπτύξουμε περαιτέρω τις σχέσεις μας και μέσω της ομάδας παρακολούθησης του Μερκοσούρ που είναι η ομάδα την οποία προεδρεύω, θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε αυτή την προσπάθεια. Να ευχαριστήσω ε, όσους βοήθησαν για την αντιπροσωπεία, την αποστολή της Αργεντινής στην Ευρωπαϊκή Ένωση, την ε, αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον Buenos Aires, τη Eurolat, φυσικά τη γραμματεία της Επιτροπής, αλλά και τις γραμματείες των πολιτικών ομάδων χωρίς την ε, ε, προσπάθεια και την εργασία τους σίγουρα δεν θα είχαμε καταφέρει να κάνουμε αυτή την αποστολή. Ευχαριστώ λοιπόν τους πάντες και ας ελπίσουμε ότι αυτή θα είναι η αρχή μιας πολύ καλής φιλίας. Ευχαριστώ πολύ. να. Πρόεδρος. Μάλιστα. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βίζας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα είμαι σύντομος γιατί τα είπε πάρα πολύ καλά ο κύριος Σάλβα να ευχαριστήσω και τη Γραμματεία για την εξαιρετική διοργάνωση και τον Πρόεδρο βεβαίως για τον ηγετικό σου ρόλο στη διάρκεια αυτής της ε, αποστολής, αυτές τις μέρες που περάσαμε μαζί στο Buenos Aires. Πιστεύω ότι είναι πολύ χρήσιμες και για τη δουλειά μας, αλλά και για να μπορέσουμε να αναπτύξουμε και δεσμούς ε, φιλίας ε, μεταξύ των μελών της Επιτροπής ΣΥΝΤΑ. Το είπατε ήδη ότι η κυβέρνηση του Πρόεδρου Μάκρη είναι πάρα πολύ ανοιχτή για να ανοίξουμε εμπορικέ σχέσει, να υπογραφεί συμφωνία με το Μερκοσούρ. Ορισμένε φορέ είχαμε την αίσθηση ότι έχουν περισσότερη δυσκολία με του γείτονέ τη ε, από πλευρά Μερκοσούρ και παρά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν είναι θέμα μόνο συμφωνία με την Ευρώπη, πρέπει να επιλύσουν και τα εσωτερικά του προβλήματα δηλαδή. Και νομίζω ότι ε, Προφανώς και υπάρχουν εκεί δυσκολίες. Είναι ε, προφανές επίσης ότι υπάρχουν κάποιες επιφυλάξεις από πλευράς βιομηχανικού τομέα. Τους ε, ανησυχεί η δύναμη της ευρωπαϊκής βιομηχανίας. Εμάς βεβαίως μας ανησυχεί η πλευρά της γεωργίας και νομίζω ότι θα πρέπει να γίνουν υποχωρήσεις κατέρωθεν. Συνοψίζοντας, νομίζω ότι αυτό που είναι σημαντικό είναι, όπως έλεγε και ο Παύλο Θάλπα, να λάβουμε συγκεκριμένες αποφάσεις. Ε, ίσως μέχρι τώρα ήμασταν μόνο σε θεωρητικό πλαίσιο και αυτό που θέλουν ε, οι Αργεντίνοι είναι να σταματήσουμε τα πολλά λόγια και να περάσουμε σε πράξεις και να κάνουμε συγκεκριμένα πράγματα ώστε να προχωρήσουν αυτές οι συμφωνίες. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Helmut Scholz στα αγγλικά. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστήσεις και από μένα στην Γραμματεία και σε όλους που εργάστηκαν παρασκηνιακά, που προετοίμασαν την επίσκεψη, πραγματικά ενδιαφέρουσα επίσκεψη. Δεν είναι πάντα εύκολο να οργανώσει κανείς πρόγραμμα που να ικανοποιεί τις επιθυμίες όλων των συμμετεχόντων. Παρόλο που ήταν σημαντική πρόκληση η ημερήσια διάταξή μας από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με διαφορετικά πράγματα ανά μισή ώρα, με συναντήσεις με πολλούς, πολλά μέλη μάλλον της κυβερνήσεως και του Κοινοβουλίου αλλά και ενδιαφερόμενα μέρη, καμιά φορά νομίζω πρέπει να σκεφτούμε και πώς μπορούμε να εμβαθύνουμε ε, στις συζητήσεις. Ομολογώ ότι για πρώτη φορά επισκέφθηκα την Αργεντινή. Ήταν σημαντικό για μένα να είμαι παρόν εκεί. Όταν μιλούμε για τη συμφωνία Μερκοσούρ, που την διαπραγματευόμαστε τώρα, αυτό σημαίνει ότι έχουμε μια χώρα, συναντήσαμε μια χώρα, και η εντύπωση μου αυτή ήταν, μπορεί να συμφωνήσουν οι συναδελφοί μου ή όχι, που είναι κατά κάποιο τρόπο η μηχανή έλξης των διαπραγματεύσεων από την πλευρά Μερκοσούρ. Είναι σημαντικό λοιπόν την στιγμή αυτή των βαθιών αλλαγών και αυτό τόνισαν όλοι ότι βρίσκονται σε φάση αλλαγής, σε μεταβατική περίοδο. Να δούμε και τι είναι πίσω από το παρασκήνιο. Είναι δηλαδή δική μας ευθύνη να δούμε και αυτούς που ήταν υπεύθυνοι στο παρελθόν για το ότι δεν προχώρησαν οι διαπραγματεύσεις ε, κόμματα της αντιπολίτευσης τα οποία εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τις ε, συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις. Δεύτερο θέμα, γιατί είπατε αρχικά, ότι βρισκόμαστε σε μια πολύ ενδιαφέρουσα φάση με την αλλαγή κυβερνήσεως στις Ηνωμένες Πολιτείες, με τι εξελίξει και σε άλλα μέρη του κόσμου αλλά και στην Ευρωπαϊκή Ένωση να δούμε ποιε είναι οι επιπτώσει του εμπορίου στι κοινωνικέ και οικονομικέ καταστάσει. Και επομένω στι διαπραγματεύσει με τι χώρε Μερκοσούρ. Ε, γνωρίζετε ότι έχουμε μια εντολή 20 ετία. Μιλούμε σε μια βάση που δεν απηχεί πλέον τις βαθιές αυτές αλλαγές που έχουν επισυμβεί και που ζούμε άλλωστε και τώρα και εδώ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και κατά πάσα πιθανότητα ισχύει αυτό και για τις χώρες εταιρού του Μερκοσούρ. Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι απαιτείται διαφάνεια, η διαπραγματευτική εντολή πρέπει να καταστεί δημόσιο κτήμα, να δούμε τι θα περιληφθούν άλλα στις διαπραγματεύσεις που ίσως έχει περιλάβει με κάποιες απλές διατυπώσεις η πρώτη διαπραγματευτική εντολή, αλλά πρέπει να δούμε τώρα τι χρειάζεται και από τη Σκοπιά, τη ζητεί και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είναι διαφορετικά τα μηνύματα που λάβαμε. και ο επικεφαλής του ομίλου Volkswagen μας ε, είπε ποια είναι η πρόκληση για την παραγωγή στην Αργεντινή που χρειάζεται μεταβατική, μακρά μεταβατική περίοδο γιατί πρέπει να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις βαθιές αλλαγές που αντιμετωπίζουν στην πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές μάλλον στην πρόσβαση στις αγορές των ευρωπαίων ανταγωνιστών. Και η ανάγκη για αυτή τη μεταβατική περίοδο υπάρχει διότι δεν προλαβαίνουν να οργανωθούν και να αντιμετωπίσουν τα ευρωπαϊκά προϊόντα. Και αυτό ισχύει και για τις κοινωνικές επιπτώσεις των διαπραγματεύσεών μας. Και από τη δική μου εμπειρία και ερμηνεύω πολλές ενδιαφέρουσες συνομιλίες με τους εταίρους μας, ότι δηλαδή οι αγροτικές επιχειρήσεις, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις από την Αργεντινή θα αποτελέσουν πρόκληση για τους Ευρωπαίους αγροτικούς παραγωγούς, ιδίως για τις μικρές και μεσαίες αγροτικές εκμεταλλεύσεις και για πολλά είδη αγροτικών προϊόντων. Και πρέπει να εξετάσουμε και το κεφάλαιο της βιωσιμότητας που είναι πάντοτε ε, εκ των όνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και πρέπει να συνδυαστεί με μια συνολικότερη επισκόπηση του τι γίνεται και ποιε είναι οι βαριές συνέπειες και στις ανθρώπινες ζωές και στην φύση των διαφόρων βιοκτώνων που χρησιμοποιούνται. Και για παράδειγμα ιδιαίτερα στην περιοχή της Πανταγωνίας και για τα προϊόντα που προέρχονται από εκεί και έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μεγάλη περιπλοκότητα των θεμάτων και από την πλευρά της αντιπροσωπείας Μερκοσούρ παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Αργεντινή και επιθυμώ να τονίσω γιατί η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα είναι κάπως προβληματικό που βλέπουμε ότι η απόφαση της κυβέρνησης για τις ταχύες πληρωμές ορισμένων οικογενειών που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα. Δεν μιλούμε μονάχα για τις επίσημες διαπραγματεύσεις. Πρέπει, με λίγα λόγια αυτό θέλω να πω, ότι πρέπει να μπούμε σε βάθος των κοινωνικών και οικονομικών εξελίξεων στην ε, χώρα αυτή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Ντάντη να ευχαριστήσω τη Γραμματεία που μας επέτρεψε να διοργανώσουμε αυτή την πάρα πολύ ε, εντατική συνεδρίαση και σε πολύ ψηλό επίπεδο ε, συνάντηση. Είχαμε και τον πρέσβη τον κύριο Σαλαφράγκα, ο οποίος είναι πρέσβης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην, κυβέρνη, ε, στην Αργεντινή. μπορέσαμε να δούμε τις αλλαγές που έχουμε στην Αργεντινή αυτή τη στιγμή και φυσικά με μεγάλες δυσκολίες όπως ε, αντιμετωπίζουν όλες οι χώρες ανά τον κόσμο που προσπαθούν να κάνουν τόσο βαθιές αλλαγές. Επίσης είδαμε μεγάλη διάθεση από πλευράς κυβέρνησης της Αργεντινής αλλά και των ε, πολιτικών δυνάμεων της Αργεντινής και σε μεγάλο βαθμό και των οικονομικών δυνάμεων της Αργεντινής να πιέσουν προκειμένου να μπορέσουμε να φτάσουμε εν ευθέτω χρόνο σε ε, μια συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση και όλη την περιοχή του Μερκοσούρ. Η Αργεντινή αυτή τη στιγμή ε, είναι η πολιτική ηγεσία του Μερκοσούρ ε, και λόγω διαστάσεων της χώρας και λόγω σημασίας της χώρας στην περιοχή του Μερκοσούρ και φυσικά αυτό το, έχουμε, το έχουν αναγνωρίσει και η κυβέρνηση της Ρουγουάης και της Παραγουάης ε, μπορέσαμε να δούμε πού βρίσκονται οι μεγάλες δυσκολίες σε μια συμφωνία σαν αυτή την οποία προσπαθούμε να συνάψουμε και υπάρχουν δυσκολίες εκατέρωθεν. Γνωρίζουμε ότι ε, σε μεγάλο βαθμό για μας αφορούν τον τομέα της γεωργίας, ε, για την Αργεντινή, αλλά νομίζω και για όλη την περιοχή του Μερκοσούρ το θέμα της βιομηχανίας και της πρόσβασης στις αγορές των ε, δημοσίων συμβάσεων πρόκειται λοιπόν για στοιχεία ε, επί των οποίων πρέπει να συνεχίσουμε τις εργασίες μας. Αλλά ενώπιον όλων αυτών των δυσκολιών ε, καταφέραμε να διαπιστώσουμε ότι όπως πολύ σωστά είπε και ο εισηγητής αλλά και είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε ότι υπάρχει διάθεση από πλευράς κυβέρνησης Αργεντινής να υπερκεράσει τα προβλήματα και να προσπαθήσει να φτάσει εγκαίρως στην επίτευξη της συμφωνίας. Επίσης, ε, μπορέσαμε να διαπιστώσαμε ότι υπάρχει και διάθεση για κάποια από τα στοιχεία κλειδί της ε, ευρωπαϊκής ε, πλευράς, παραδείγματος χάρη τις γεωγραφικές ενδείξεις. Πρόκειται για ένα θέμα για τη γεωργία μας. Δεν ολοκληρώθηκε, αλλά υπάρχει ανάγκη να εμβαθύνουμε και υπάρχει διάθεση από ό,τι βλέπουμε να αναγνωριστούν. Οι ε, χρόνοι επίσης της ανταλλαγής προσφορών είναι πολύ ε, μεγάλη στο χρονοδιάγραμμα που παρουσίασε η Γεργεντινή. 15 χρόνια ε, διαπιστώσαμε ότι υπάρχει διάθεση ε, να μειώσουμε λοιπόν αυτό το μεταβατικό διάστημα. Τα περισσότερα στοιχεία της αποστολής ε, τα είπε και ο εισηγητής, τα είπατε και εσείς κύριε Πρόεδρε και οι προλαλήσαντες. Εγώ λοιπόν θα ήθελα απλώς, ε, ολοκληρώνοντας την παρέμβασή μου, να πω ότι πρόκειται για στρατηγική εμπορική συμφωνία και πρέπει να την επισημάνουμε τη στρατηγική πτυχή. Και δεδομένου ότι σήμερα το πρωί ξυπνήσαμε ή περάσαμε τη νύχτα ενώπιον της τηλεοπτικής οθόνης ε, παρακολουθώντας τα αποτελέσματα των Αμερικανικών εκλογών, η στρατηγική σημασία αυτής της συμφωνίας είναι ακόμα μεγαλύτερη. Γι' αυτό λοιπόν πιστεύω κύριε Πρόεδρε και συνάδελφοι ότι πρέπει ε, να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε αυτή τη συμφωνία, να βοηθήσουμε αυτή τη διαπραγμάτευση, προσπαθώντας να βρούμε σημεία συμβιβασμού, ε, τα οποία να μας επιτρέψουμε εγκαίρως να καταλήξουμε σε μια συμφωνία, ώστε η Ευρωπαϊκή Ένωση να ε, συνεργαστεί με μια ε, περιοχή με την οποία είναι συνδεδεμένη από ιστορικής, οικονομικής πλευράς, από πλευράς αξιών και θα αποτελέσει και ένα πολύ σημαντικό εμπορικό εταίρο για όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. E, Ευχαριστώ αγαπητέ Πρόεδρε. Νομίζω ότι λέχθηκαν σχεδόν όλα. Θέλω μόνο να πω ότι μετά την νύχτα που μας πέρασε, δηλαδή ενώ τις αμερικανικές εκλογές, δεν έχω τίποτα θετικό να πω. Είχα αποφασίσει μάλιστα να μην μιλήσω. Το ταξίδι ήταν θαυμάσιο οργανωμένο πάντω και ομολογώ ότι είμαι ιδιαίτερα ικανοποιημένος από τις προπαρασκευαστικές εργασίες και όπως έγιναν. Εγώ χαίρομαι για τις ε, συναντήσεις οι οποίες έρχονται να επιβεβαιώσουν τα όσα γνωρίζαμε ήδη εκ των προτέρων και νομίζω ότι οι σχέσεις μας με την χώρα αυτή είναι εξαιρετικέ. Εάν υλοποιηθούν όλα όσα επιθυμεί η κυβέρνηση Αργεντινής, νομίζω ότι η χώρα αυτή θα παίξει ένα πολύ σημαντικό ρόλο και θα έχει ένα πολύ θετικό μέλλον στην περιοχή αυτή. Άκουσα πολύ αισιοδοξία από τα λόγια των συναδέλφων μου. Δεν είμαι τόσο αισιόδοξο ε, όσο οι συναδελφοί μου, σε αυτό, αυτό να με έχει επηρεάσει η νύχτα, η οποία, ε, πώς να πω, συρρήκνωσε κάπως την αισιοδοξία μου. Και στην Αργεντινή γίνονται εκλογέ του χρόνου. Η κυβέρνηση που έχουν τώρα εκεί και που ασκεί θαυμάσια το κυβερνητικό έργο δεν ξέρουμε αν θα διατηρήσει την εξουσία. Δεν ξέρουμε αν έχει μέλλον. Αυτό σημαίνει ότι η συμφωνία θα πάρει χρόνια με τις διαπραγματεύσεις και μέχρι ό,τι υλοποιηθεί Έχουμε χρόνο ακόμη. Βεβαίως, πράγματι θα είναι σημαντική η πρόκληση, έχετε δίκιο σε αυτό. Νομίζω όμως ότι η στρατηγική σημασία της συμφωνίας αυτής και ειδικώ εν ώψη των αποτελεσμάτων των Αμερικανικών εκλογών είναι σημαντική, η σημασία είναι μεγάλη. Θα παρακολουθήσουμε άλλωστε ενεργά τη διαδικασία αυτή. Ευχαριστώ. Εδώ λίγη συζήτηση για το θέμα αυτό της ημερησίας διάταξης και το υπαριθμόν 6. Πρόκειται για ανταλλαγή αλληλογραφίας μεταξύ Βραζιλίας και Ευρωπαϊκής Ένωσης για ρυθμίσεις του ΠΟΕ σχετικά με την ένταξη της Κροατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Διαδικασία η οποία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί. Το Συμβούλιο χρειάζεται κάποιο διάστημα ακόμη για να κάνει τις σχετικές επαληθεύσεις. Θα μας τα πει αυτά όμως ο μόνιμος συγκητής μας για το Μερκοσούρ, ο κ. Σάλβα. Ε, Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, δεν είναι η πρώτη έκθεση της Επιτροπής μας για την προσαρμογή συμφωνιών με τρίτες χώρες ε, λόγω της προσχώρησης της Κροατίας. Με την ε, προσχώρηση αυτή διευρύνθηκε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όπως και στις ε, προηγούμενες περιπτώσεις βεβαίως, ε, όπως είναι διατυπωμένα τα άρθρα 24 και 6 της ε, συμφωνίας ε, ΓΚΑΤ, ε, της Γενικής Συμφωνίας Δασμών και Εμπορίου και το άρθρο 27, αυτή η διαδικασία την οποία ξεκινούμε να συζητούμε σήμερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στόχο έχει να εγκρίνει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μία συμφωνία που θα ολοκληρώσει τις διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ε, Μερκοσούρ για την συνεννόηση που πρέπει να υπάρχει όπως καθορίζει ο ΠΟΕ όταν ένα κράτος μέλος το οποίο ε, συμμετέχει σε μία τελωνιακή ένωση σκοπεύει ε, να αυξήσει τα δικαιώματα τα οποία απορρέουν από τη συμφωνία. Η Επιτροπή έκανε διαπραγματεύσεις και προσπαθούν να έχουν μια αντισταθμιστική προσαρμογή η οποία θα είναι ικανοποιητική και θα λαμβάνει υπόψη της τις ε, μειώσεις ε, των δασμών ε, και των δικαιωμάτων. Ε, προφανώς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα δώσει τη σύμφωνη γνώμη του για την οριστικοποίηση τη συμφωνίας μεταξύ Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Ομοσπονδιακή Δημοκρατία τη Βραζιλία, διότι λόγω της διεύρυνσης της Τελωνιακής Ένωσης μετά την προσχώρηση της Κροατίας και βάσει και των κανόνων του ΠΟΕ, πρέπει να εξετάσουμε μια πιθανή αντισταθμιστική προσαρμογή του ε, δασμολογικού καθεστώτος που ισχύει αυτή τη στιγμή. Πιο συγκεκριμένα, θα ήθελα να σας αναλύσω λίγο καλύτερα την υπόθεση αυτή. Ε, όπως και σε προηγούμενες περιπτώσεις ε, με άλλους εταίρους, ε, αντιλαμβάνουμε ότι υπάρχουν κάποιοι τομείς που πλήττονται ε, ή επηρεάζονται περισσότερο από αυτές τις προσαρμογές. Γι' αυτό λοιπόν ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και κυρίως τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου και τη Γενική Διεύθυνση Γεωργίας για αυτή την πρώτη ανταλλαγή απόψεων και θέλουμε να μας εξηγήσουν αναλυτικά τη διαδικασία που ακολουθείτε για τον υπολογισμό των παραχωρήσεων που καθορίζονται από τον ΠΟΕ. Ε, υπάρχουν κάποια θέματα τα οποία αφορούν το τομέα της ζάχαρης, για παράδειγμα, ή των ε, πουλερικών. Ε, ήρθαν σε επαφή με εμά οι σχετικοί κλάδοι, γι' αυτό λοιπόν θα θέλαμε να ξέρουμε τι μπορεί να μας πει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από αυτού. Ε, αυτή η ανταλλαγή απόψεων θα μας βοηθήσει να εκπονήσουμε μια έκθεση η οποία θα αποτελέσει και σύσταση για την έγκριση της συμφωνίας. Αυτή τη στιγμή βεβαίως και το Συμβούλιο μας διαβιβάσει την επίσημη συμφωνία πριν φυσικά τεθεί σε εφαρμογή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Ντάντης και ο συζητητής. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο εισηγητής έκανε μια πολύ σαφή παρουσίαση της συμφωνίας που συζητούμε σήμερα. Νομίζω ότι η μεγαλύτερη δυσκολία και το μεγαλύτερο πρόβλημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η δυνατότητα να υπάρχει ένας δασμός για έξι ε, χρόνια σε ένα πολύ καλό ποσοστό για το τομέα της ζάχαρης από πλευράς Βραζιλίας ε, και κυρίως ε, για τα ζαχαροκάλαμα τα οποία προορίζονται για επεξεργασία. Θα υπάρχει 11 ευρώ ανασέντ και να φτάσουμε μετά ε, στη συνέχεια στα 98 ε, ευρώ από την 8η χρονιά. Ε, είναι 78.000 τόνοι η ζάχαρη που μας ενδιαφέρει. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι κατά πάσα πιθανότητα θα υπάρχουν συνέπειες σε σχέση με αυτά τα οποία εξάγονταν από τη Βραζιλία στην Κροατία στο παρελθόν. Θα πρέπει όμως να δούμε πώς, ε, ε, τι σχέση έχει αυτό με το παρελθόν ο αριθμός αυτός των τόνων. Θα πρέπει λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας πει τι ποσοστά ε, εξάγονταν ε, στο παρελθόν από τη Βραζιλία στην Κροατία. Να δούμε κατά πόσον αυτές οι ποσότητες είναι αναλογικές σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια για τις εξαγωγές της Βραζιλίας προς την Κροατία. Ευχαριστώ κύριο Τσάρντιλ. πολύ σύντομα. Είναι μια κανονική διαδικασία. Κάναμε το ίδιο στις προηγούμενες διευρύνσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. έτσι ώστε μια θεωρούμενη ως τυπική διαδικασία ως ομάδα δεν μπορούμε παρά να είμαστε υπέρ μιας τέτοιας διαδικασίας είναι καλό να γνωρίζουμε ποια προϊόντα θα καλύπτονται από αυτήν. Αλλά δεν νομίζω ότι το ζήτημα είναι αμφιλεγόμενο ή ότι πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο κάποια τροποποίηση ή περαιτέρω συζητήσει. Είμαστε εντάξει με αυτό. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Τσαράτσονοβα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίση να ευχαριστήσω τον εισηγητή για την παρουσίασή του. Υποστηρίζω τα σχόλιά του σε γενικές γραμμές. Αλλά με αυτή την ευκαιρία θα ήθελα να τονίσω αυτό που όλοι μας γνωρίζουμε, πως η ε, πως η Βραζιλία αποτελεί την σημαντικότερη αγορά για τους εξαγωγείς και τους επενδυτές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και η Βραζιλία στρέφεται προς την απελευθέρωση της αγοράς της η Βραζιλία εφαρμόζει τελευταία διάφορα μέτρα περιορισμού της αγοράς σε διάφορους τομείς. Γι' αυτό και θα ήθελα να ενθαρρύνω τον Επίτροπο να συνεχίσει να ασκεί πίεση στην Βραζιλία ως προς αυτό. Επίσης, στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μέρκοσου πρέπει να επιταχύνουμε και να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία για να επιτύχουμε στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων αυτών ένα αποτέλεσμα. Χέλμουτ. Ευχαριστώ. Και εγώ θα ήθελα να υποδείξω πρώτα απ' όλα ευχαριστώ και εγώ τους συζητητές πως πρέπει να παρατηρήσουμε, να θεωρήσουμε το ερώτημα αυτό επίσης στις περίπλοκες διαστάσεις που έχουν οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Eurosur, Mercosur, συγγνώμη. Κάποια προβλήματα συνδέονται με το ότι έχουμε εντελώς διαφορετικές αφετηρίες σήμερα και έχουμε να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά αποτελέσματα και πρέπει να βρούμε λύσεις γι' αυτό. Παραδείγματος χάρη εισαγωγέ ζάχαρης από την Κροατία στην Κροατία από τη Βραζιλία σχετίζεται με την αποχώρηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης από τη βραζιλιάνικη αγορά ζάχαρης. Δηλαδή έχουμε δηλαδή οι λύσεις που θα επιτύχουμε δεν πρέπει να γίνονται εις βάρος μιας δίκαιης φιλικής προς το περιβάλλον εμπορικής πολιτικής πρέπει να συνεννοηθούμε ως προς το θεματικό πεδίο αυτό. Τι σημαίνει για τους Βραζιλιάνους παραγωγούς, για τις θέσεις εργασίας και για το ζήτημα των κοινωνικών και περιβαλλοντικών προτύπων εκεί και για τη δυνατότητα της εγχώριας παραγωγής. Εδώ πιστεύω πως πρέπει να συνεχίσουμε να παρακολουθούμε από κοινού με τον εισηγητή και να συζητήσουμε με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς, για το πώς μπορούμε να βρούμε μία λύση για την πρόκληση αυτή. Ευχαριστώ κυρία Μπιγκίν. Ευχαριστώ. Εμείς, των πέντε αστέρων δηλαδή, και εγώ προσωπικά, Δεν έχω να πω τίποτε γιατί δεν είναι παρόν ο αρμόδιος συνάδελφός μου. Ακολουθούν άλλοι συναδελφοί. Ε, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, με συγχωρείτε. Ευχαριστώ και καλημέρα. Κυρίε και κύριοι ευρωβουλευτέ, λέγομαι Μπέντφορντ, είμαι επικεφαλή τμήματο για θέματα ΠΟΕ στην αρμόδια Γενική Διεύθυνση τη Κομισιόν και ήμουν επικεφαλή των διαπραγματεύσεων για το θέμα αυτό που συζητείτε σήμερα. Πρώτα, θα συμφωνήσω με τον εισηγητή σε ό,τι αφορά την περιγραφή της καταστάσεως. Πρόκειται για το τρίτο σχέδιο συμφωνίας, το οποίο τίθεται υπόψη της Επιτροπής σας ως αποτέλεσμα της ε, κουρατικής εντάξεως και για τα άρθρα 24.6 και 26 του ε, ε, ΓΑΤ. Έχει την νομική υποχρέωση η Ευρωπαϊκή Ένωση υπό την ισχύ των διατάξεων του ΠΟΕ να φροντίσει ώστε οι συνθήκες πρόσβασης στην αγορά της ε, Ευρώπης των 28 να είναι ισότιμες με αυτές που ίσχυαν για την Ευρώπη των 27 και για την Κροατία προ της εντάξεως. Αυτό είναι το βασικό. Δηλαδή να διασφαλίσουμε ότι η κροατική ένταξη δεν επιδεινώνει την πρόσβαση στις ευρωπαϊκές αγορές για άλλες χώρες που είναι και αυτές μέλη του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου. και σε διαπραγμάτευση μπαίνουν προϊόντα όπου οι δασμοί, οι κρατικοί δασμοί ήταν χαμηλότεροι από αυτούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, διότι όταν εντάσσεται η Κροατία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, υιοθετεί τους δασμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις περιπτώσεις όπου σημειώνεται λοιπόν αύξηση των δασμών, των εισαγωγικών δασμών, πρέπει να διαπραγματευτούμε με τους βασικούς προμηθευτές, μέλη του ΠΟΕ, και να διαπραγματευτούμε κάποια αντιστάθμιση, ώστε η κατάσταση να επανέλθει στην αρχική, για αυτούς δηλαδή, πριν από την ένταξη. Στην περίπτωση τη Βραζιλίας, δύο κυρίω προϊόντα προμήθευε η Βραζιλία, που εντάσσονται στο σχέδιο συμφωνία που έχετε μπροστά σας σήμερα, ζάχαρη και πουλερικά, μεταξύ αυτών και κρέα γαλοπούλας. Και στι δύο περιπτώσει αυτέ η κροατική δασμή ήταν χαμηλότερη από τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα χρειάζεται να δώσουμε αντιστάθμιση. Θα αναφερθώ πρώτα στο κρέας πουλερικών. Εκεί η κροατική δασμή ήταν πολύ χαμηλότερη από τους ευρωπαϊκούς. Όταν λοιπόν υιοθετήσει τους ευρωπαϊκούς δασμούς, αυτή είναι σχεδόν απογορευτική. Είναι αδύνατον δηλαδή να γίνουν εισαγωγέ σε απογορευτικό, με απογορευτικού τέτοιου δασμού. Άρα πρέπει να δώσουμε λοιπόν αντιστάθμιση για το ποσό αυτό που εισήγει η Κροατία. Παίρνουμε λοιπόν το μέσο όρο τριών ετών πριν από την ένταξη, σημειώνουμε αυτόν τον όγκο εισαγωγών και αυτόν και για αυτόν χρωστούμε αντιστάθμιση. Και ο όγκος αυτός θα ήταν περίπου 6.500 τόνοι ε, πουλερικών και ε, περίπου 1.500 τόνοι ε, κρέατος γαλοπούλας. Δίνουμε λοιπόν όχι βέβαια απεριόριστη παραχώρηση, γιατί αυτή, ε, αυτό ισχύει για την Κροατία τότε. Δηλαδή μπορούσαν να εισάγουν, να εισάγουν μάλλον όσο κρέας πλευικών και γαλοπούλας ήθελαν. Τώρα όμως εμείς βάζουμε αυτό το όριο. 6.500 τόνους πουλερικών και 1.200 γαλοπούλες Βάζουμε λοιπόν αυτό τον περιορισμό. Και εκεί ο δασμός μπαίνει στο 0. Δηλαδή είναι σχετικά μικρό το ποσό σε σύγκριση με αυτό που εισάγει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν αναμένουμε λοιπόν να είναι πολύ μεγάλο το αποτέλεσμα. Για τη ζάχαρη η κατάσταση είναι λίγο πιο περίπλοκη. Η Κροατία είχε δασμό χαμηλότερο, αλλά αυτόνομα η Κροατία επέβαλε για μια επταετία πριν από την ένταξη ακόμα χαμηλότερα. Πάντοτε υπό την ισχύ των διατάξεων του ΠΟΕ μπορεί να το κάνει κανεί αυτό. Μπορεί να επιβάλλει δηλαδή ακόμα χαμηλότερο δασμό και αυτό έκανε η Κροατία η κατάσταση είναι περίπλοκη και θα έλεγα μάλιστα μοναδική. Δεν έχουμε ξανασυναντήσει τέτοια κατάσταση σε παρόμοιε διαπραγματεύσει. Ακολουθήσαμε του ίδιου κανόνε, εξετάσαμε δηλαδή τον όγκο των εισαγωγών στην Κροατία πριν από την ένταξη και αυτή είναι η βάση των όγκων εισαγωγή 114.000 τόνοι που εισήχθησαν στην ε, Κροατία πριν από την ένταξη και αυτή είναι η βάση για τις αντισταθμίσεις που χορηγούμε τώρα. Το χωρίσαμε 78.000 τον για τη Βραζιλία και 78.000 που είναι ανοιχτοί για όλες τις εισαγωγές. Και αυτό απηχεί την κατάσταση της Κροατίας πριν από την ένταξη. Κάποιες από τις εισαγωγές αυτές γίνονταν ειδικά από την Βραζιλία και άλλες ήταν πάλι ανοιχτός ο εκεί για ε, εισαγωγές από άλλες χώρες. Ζάχαρης πάντα. 114.000 τόνοι ζάχαρης δεν είναι και καμιά αμεληταία ποσότητα. Ήταν λοιπόν σκληρέ οι διαπραγματεύσει. Εν τέλει, καταλήξαμε σε μια συμφωνία που απηχεί με μεγάλη ακρίβεια τους κανόνες του ΠΟΕ για τον όγκο αντιστάθμισης που πρέπει να δώσουμε. Δεν δίνουμε παραπάνω από αυτό που θεωρούμε ότι είμαστε απολύτως υποχρεωμένοι σύμφωνα με τους κανόνες του ΠΟΕ. Μια από τις καταστάσεις που χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε ήταν και το γεγονός ότι η Κροατία εφήρμοζε αυτό τον αυτόνομο δασμό, πάρα πολύ χαμηλό, για μια επταετία και καταλήξαμε σε μια συμφωνία με τους Βραζιλιάνους ότι τελικά για μια περίοδο 7 ετών μετά από την ένταξη, μετά από εδώ τη συμφωνία, θα δώσουμε ένα παρόμοιο αυτόνομο καθεστώς. Το ίδιο λοιπόν προσωρινό χαμηλό καθεστώς μετά από την αρχή εφαρμογή συμφωνία. Έξι χρόνια δηλαδή, χαμηλότερα, μετά ένα χρόνο θα αυξηθεί και μετά θα έρθει στο κανονικό δασμό που είναι 98 ευρώ τον τόνο. Για να σας εξηγήσω λοιπόν την ασύνηθη αυτή κατάσταση που δεν έχουμε ξανακάνει τέτοιο πράγμα, δεν έχουμε ξαναδεί δηλαδή τέτοια κατάσταση ε, όπως αυτή τη διαπραγματεύση. Η διαπραγμάτευση ήταν και κεντρικό στοιχείο για να κρατήσουμε τους όγκους σε αυτό το επίπεδο που τους κρατήσαμε, διότι ζητούσαν για πολύ περισσότερο, ζητούσαν 320.000 τόνους. Καταφέραμε λοιπόν να τους κατεβάσουμε στο 1 τρίτο του όγκου αυτού, διατηρήσαμε λοιπόν το ελάχιστο αυτό, με ένα προσωρινό χαμηλότερο δασμό για την περίοδο των 7 ετών. και οι συναδελφοί που είναι αρμόδιοι για την αγορά της ζάχαρης ε, μας επιβεβαιώσαν ότι ήταν προς το συμφέρον μας να κρατήσουμε τον όγκο των εισαγωγών στο χαμηλότερο δυνατό επίπεδο. Και αυτό ήταν στο επέκεντρο των διαπραγματεύσεων μας. Ελπίζω ότι σχετικά, με σχετική συντομία μπόρεσα να σας εξηγήσω τα στοιχεία μιας περίπλοκης διαπραγμάτευσης και ευχαρίστω να απαντήσω σε ερωτήσεις που ίσως έχετε. Ευχαριστώ. Εσεί κύριε Σιγητά πάλι. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τι ε, διεξοδικότατε εξηγήσει. και όπω είπαν και οι συνάδελφοι, του οποίου σα ευχαριστώ, αυτή είναι μία από τι συνηθισμένε διαδικασίε και ελπίζω με το επικοδομητικό πνεύμα που επέδειξαν να μπορέσουμε να προχωρήσουμε όσο το δυνατόν πιο εύκολα. Δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Ευχαριστώ για τη συνεισφορά σας και θα συνεχίσουμε τις εργασίες. Ευχαριστώ πολύ. Ο μόνιμος εισηγητής θα εκπονήσει ένα σχέδιο έκθεσης και με αυτή τη βάση μπορούμε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Οπότε κλείνω το σημείο 6 της ημερήσιας διάταξης, προχωρούμε στο 7, το οποίο όπως είπαμε μετατέθηκε, περνάμε στο 8 δηλαδή. Το ζήτημα εδώ είναι, το θέμα είναι το φινικέλαιο και η αποψήλωση τροπικών βαστών. Έχουμε μια τοποθέτηση για μια έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, αλλά υπό το πρίσμα του γεγονότος πως η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εισαγωγέας φινικελαίου σε παγκόσμιο επίπεδο με 7 εκατομμύρια τόνους ανά έτος. Έχουμε πολλές συνέπειες για το, για το εμπόριο. Έχουμε και κάποιες εμπορικές συμφωνίες με σχετικές χώρες όπου το ζήτημα του κανονισμού Φλακτ και εθελοντικών εμπορικών συμφωνιών παίζουν επίσης σημαντικό ρόλο για την βελτίωση της βιωσιμότητας. Οπότε δίνω το λόγο στην εισηγήτριά μας, την κυρία Μπιγκίν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, όπως όλοι γνωρίζετε, το φινικέλαιο είναι ένα προϊόν στο επίκεντρο ε, πολλών συζητήσεων στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και ανησυχίας ε, από πλευράς Ευρωπαίων πολιτών και δικαίως, διότι υπάρχουν και κίνδυνοι για την υγεία, αλλά και περιβαλλοντικές ε, ε, ζημίες. Ε, συζητήσαμε πάρα πολύ τα θέματα υγείας και περιβάλλοντος που σχετίζονται με το έλαιο. Ε, δεν έχουμε πει όμως πολλά για την προέλευσή του, για τη χρήση του και για την εμπορική πλευρά αυτού του τόσο επιζήμιου προϊόντος. Το φινικέλαιο από μόνο του είναι το 40% του παγκοσμίου εμπορίου σε φυτικά έλαια. 7 εκατομμύρια τόνους το χρόνο ε, έρχονται στην Ευρωπαϊκή Ένωση, κυρίως από τη Μαλαισία και την Ινδονησία, που είναι και η μεγαλύτερη παγκόσμια παραγωγή, διότι μαζί αποτελούν το 85 με 90% της παγκόσμιας παραγωγής. Πολλές ε, διατροφικές βέβαια βιομηχανίες μειώνουν τη χρήση φενικελαίου, κυρίως ε, για λόγους διαφήμισης. Πολλοί κόσμος όμως δεν γνωρίζει ότι το φενικέλαιο χρησιμοποιείται και για την παραγωγή βιοντίζελ και επίσης ε, η χρήση του για την παραγωγή βιοκαυσίμων κατά πάσα πιθανότητα θα αυξηθεί ε, λόγω της μείωσης της ζήτησης ε, για διατροφικά προϊόντα. Επομένως, η αυξημένη ζήτηση φινικελαίου δημιουργεί μεγάλες πιέσεις στο περιβάλλον για την βιοπικιλότητα των ζώων και των φυτών λόγω της αποψήλωσης των δασών. Πρέπει λοιπόν να μειωθεί η χρήση του προϊόντος και να δώσουμε κίνητρα από την άλλη πλευρά για την βιώσιμη παραγωγή του. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο δεύτερος εισαγωγέα παγκοσμίων σε αυτού του προϊόντο. Εισάγουμε, επαναλαμβάνω, 7 εκατομμύρια τόνου το χρόνο. Επομένως, εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι βρισκόμαστε σε θέση να υπαγορεύσουμε τους κανόνες του παιχνιδιού. Στην γνωμοδότηση, στην οποία είμαι συντάκτηρια εδώ στην Επιτροπή, θέλω να προτείνω την ε, τον καθορισμό διαφορετικών ε, ποσοστών ε, για το φινικέλαιο και να ζητήσουμε να υπάρχουν ποσοστώσεις ε, με βάση και τη βιώσιμη παραγωγή. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και πώς γίνεται το φινικέλαιο να μην είναι στις μηδενικές ποσοστώσεις όσον αφορά τους δασμούς. Ε, Επίση, να πω ότι η παραγωγή για το βιοδίζελ θα πρέπει να είναι βιώσιμη και να υπάρχει και κατάλληλη ε, επισήμανση εάν τα βιοδίζελ παράγονται με χρήση φινικελαίου. Ελπίζω να σας παρασίασα τα βασικά μου επιχειρήματα. Ε, θα κάνω ό,τι μπορώ φυσικά και θα συνεργαστώ με τους κοιόδη συντράκτε για να μπορέσουμε να έχουμε και μια πολύ καλή γνωμοδότηση και μια κοινή άποψη για αυτό το θέμα το οποίο είναι πάρα πολύ ε, σημαντικό. Ευχαριστώ πολύ στον Σκιώδη κύριο Βίνκλερ, ο λόγος. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Αγαπητέ συναδελφέ, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Φυσικά και πιστεύω πως ένα σημαντικό ζήτημα είναι ο αντίκτυπος και οι επιπτώσεις για τις τοπικές κοινότητες και το τοπικό περιβάλλον, που δεν είναι πάντα ένα ισορροπημένο φαινόμενο, αλλά πρέπει να έχουμε κατά νου ένα βιώσιμο τρόπο προς τα μπροστά, για να συνδυασούμε την οικονομική ανάπτυξη και την δημιουργία θέσεων εργασίας με τις, με τις κοινωνικές και περιβαλλοντικές διαστάσεις. Ένας πιθανός δρόμος μπροστά μπροστά θα μπορούσε να είναι το, το σχέδιο πιστοποίησης φινικελαίου που ήδη έχουμε και τέλος πιστεύω πως ήδη έχουμε πολύτιμες εμπειρίες, ιδίως με τα ορυκτά συγκρούσεων, στην αντιμετώπιση ζητημάτων ανάπτυξης, κοινωνικών και κοινοτικών ζητημάτων και εμπορίου και των αναγκών μας ως οικονομικό μπλοκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Αν βρούμε την κατάλληλη ισορροπία, τότε βρισκόμαστε σε καλό δρόμο. Ευχαριστώ πολύ για την εργασία σας και για τη συνεργασία σας. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Τσάλη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, μιλώ εκ μέρους του κυρίου Καμάλ που είναι ο σκιώδης εισηγητής. Δυστυχώς δεν βρίσκεται εδώ επί του παρόντος και οπότε γνωρίζετε είναι επίσης μόνιμος εισηγητής για την εμπορική συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Μαλαισίας. Όσον αφού έχουμε το ζήτημα των παραβιάσεων των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που συνοδεύουν το ζήτημα αυτό, αλλά αυτό που ήθελα να πω είναι, αναφέρεται στην βιώσιμη ανάπτυξη. Το, για το βιώσιμο φινικέλαιο θα θέλαμε να εκφράσουμε την υποστήριξή μας. Αλλά ωστόσο υπάρχουν πολλά εμπόδια ακόμα για την βιώσιμη παραγωγή φινικελαίου και θα θέλαμε να τονίσουμε προς συζήτηση κυρίως τρία σημεία. Πρώτον, αν και σημειώθηκε πρόοδος στο ζήτημα του όγκου και της ποικιλία του πιστοποιημένου φινικελαίου, αυτό ισχύει μόνο για τα κύρια παράγωγα και για τα λιγότερο σημαντικά φινικέλαια, ιδίω σε τομεί πέραν του τομέα των τροφίμων, απομένουν πολλά που πρέπει να γίνουν. Δυστυχώ υπάρχουν ασυνέχειε όσον αφορά ίσονα παράγωγα που χρησιμοποιούνται παραδείγματο χάρη για οικιακή χρήση. Θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην ετικετοποίηση καθώς έχουμε ασυνεχεία στη διατροφική αλυσίδα. Δεύτερον, πρέπει να δημιουργήσουμε διαχωρισμένες εφοδιαστικές αλυσίδες. Αλλά η ταχύτητα του φαινομένου δεν μας επέτρεψε να καταρτήσουμε αρκετές εφοδιαστικές αλυσίδες. Και τέλος πρέπει να γίνουν πολύ περισσότερα ακόμα για να ληφθούν υπόψη οι μικροί παίκτες στην εφοδιαστική αλυσίδα. Πολύ μικροί προμήθευτες αντιμετωπίζουν το πρόβλημα ότι είναι απαγορευτικό το κόστος της διαπίστευσης και της πιστοποίησης και αυτό τους εξωθεί έξω από την αγορά. Ως συμπέρασμα, λίγες λέξεις σχετικά με το σύμφωνο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαλαισίας. Συζητήσεις όπως αυτές καθιστούν, δείχνουν πόσο επιτακτική είναι η ανάγκη να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Δεσμευόμαστε για την προστασία των φυσικών πόρων και την βιώσιμη χρήση των εκμεταλλεύσιμων πόρων. Πρέπει να διασφαλίσουμε πως το εμπόριο δεν θα καταλήξει σε καταστροφή προστατευόμενων περιοχών. Αυτό ήταν. Ευχαριστώ πάρα πολύ εκ μέρους του κύριου Καβάλ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Σούστερ. Ευχαριστώ πολύ καθώς η σκιώδης συγκίτριά μας δεν μπόρεσε να έρθει, με παρακάλεσε να διαβάσω την τοποθέτησή της, την γνωμοδότησή της. Αγαπητοί συνάδελφοι, το φινικέλιο βρίσκεται παντού στα τρόφιμά μας, στα απορριπαντικά μας, αποτελεί πηγή τεράστιων κερδών για πολυεθνικούς οργανισμούς, ενώ καταστρέφει το βίος μικρών νοικοκυριών. Έχουμε το πρόβλημα της αποψήλωσης της απώλειας βιοπικιλότητας ως αποτέλεσμα της κατανάλωσης φινικελαίου. 66 εκατομμύρια τόνοι ετησίως είναι η παραγωγή του που το κάνει το πιο το φυτικό έλαιο που παράγεται περισσότερο. Τόσο στην Αφρική όσο και στην Ασία έχουμε εκπομπή τεράστιων ποσοτήτων διοξιδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα λόγω της παραγωγής του. Η Ινδία θα προσπεράσει το 2015 τις Ηνωμένε Πολιτείε όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα. Στην Ινδονησία έχουμε χιλιάδες συγκρούσεις σε σχέση με το διοικησιακό καθεστώς γεών που σχετίζονται με το φινικέλαιο. Έχουμε επίσης συγκρούσεις ε, ακόμη και σε υποτιθέμενα οικολογικές θητείες. Τι μπορούμε να κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Πρέπει να ασκήσουμε πίεση για τη σύναψη εμπορικών συμφωνιών οι οποίες θα θα περιέχουν κεφάλαια περί βιώσιμης ανάπτυξης τα οποία θα πρέπει να εστιάζουν στα ανθρώπινα δικαιώματα, στο περιβάλλον και στη βιοπικιλότητα. Επίσης πρέπει να λάβουμε κατάλληλα μέτρα για αντιμετώπιση και πρόληψης της αποψήλωσης. Πρέπει να πολεμήσουμε ενάντια στην εκμετάλλευση των εργατών και των παιδιών. Πρέπει να ασχίσουμε πίεση στις εταιρείε να εφαρμόσουν κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα κατά την παραγωγή φινικελαίου το οποίο θα πρέπει να παράγεται με πιο ηθικό τρόπο. Η διαφάνεια και η χνηλασιμότητα είναι σημαντικά στοιχεία γι' αυτό. Στο τέλος της ημέρας οι εταιρείε του τομέα παραγωγής φινικελίου πρέπει να δεσμευτούν πως το, η παραγωγή τους είναι βιώσιμη για το περιβάλλον, την βιοπικιλότητα, αλλά προσφέρει επίσης δίκαιες συνθήκες για τους καλλιεργητές και πως δεν βασίζεται στην, αναγκαστική παιδική εργασία. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρος. Ευχαριστώ πολύ. Τώρα για το Άλντε, η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα επίσης να ευχαριστήσω τον εισηγητή, την εισηγήτρια για την εισαγωγή της και τα προκατακτικά της σχόλια για αυτό το πολύ σημαντικό και πολιτικά ευαίσθητο θέμα. Η εξέλιξη του φινικελαίου προκάλεσε την καταστροφή τροπικών δασών, το οποίο αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα οικολογικά προβλήματα στον πλανήτη μας πριν από 30 χρόνια είχαμε 1500 εκατομμύρια εκταρίων ε, για την καλλιέργεια φινικελαίου. Αυτό έχει εκατονταπλασιαστεί υπερβαίνοντας πλέον το μέγεθος της χώρας μου, της τσεχικής δημοκρατίας. Οι συνέπειες της παραγωγής φινικελαίου πολλές φορές περιλαμβάνουν την επιδείνωση του περιβάλλοντος χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή του μολύνουν σε μεγάλο βαθμό το περιβάλλον με επιπτώσεις τόσο για τους ανθρώπους όσο και για την πανίδα. Δεδομένων των γεγονότων αυτών, πιστεύω πως πρέπει να καταστήσουμε σαφές τους εμπορικούς εταίριους μας για τους κινδύνους που ενέχει η υπερμέτρη χρήση φινικελαίου σε, σε τρόφιμα και σε προϊόντα πέραν των τροφίμων. Αυτό δεν σημαίνει πως στρεφόμαστε κατά της παραγωγής, αλλά πως η παραγωγή πρέπει να γίνει πιο υπευθυνή. Πιστοποιητικά βιώσιμου φινικελαίου είναι ένας τρόπος αντιμετώπισης του ζητήματος. Επίσης πρέπει να σκεφτούμε πώς μπορούμε να ενημερώσουμε καλύτερα τους καταναλωτές για τη χρήση φινικελαίου προσμένω το, το σχέδιο της εισηγήτριας για το ζήτημα αυτό και τη συζήτηση με τους άλλους εμπλεκόμενους. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Το Γκούε, Χέλμουτ. Ευχαριστώ πολύ, Χέλμουτ. Και ο δικός μας Κιώδης δεν είναι εδώ. Οπότε μου ζήτησε να διαβάσω εγώ την θέση του Γκούε. Εν γέννη, συμμεριζόμαστε την γραμμή της εισηγήτριας όσον αφορά την πιστοποίηση σχετικά με ζητήματα των τροπικών δασών. Το φινικέλαιο μαζί με την εξόριξη κάποιων ορυκτών αποτελεί έναν από τους κύριους λόγους για την αποψήλωση τροπικών δασών. Μόνο η Ινδονησία και η Μαλαισία παράγουν 85% του παγκόσμιου φινικελαίου. Στην Ινδονησία, παραδείγματο χάρη, ευθύνεται για 75% τη αποψήλωση σε κάποιες περιοχές του Μπόρνεο. Η εμπορία παραγόγων φινικελαίου αποτελεί αιτία επίσης για παραχώρηση πολύ μεγάλων γεών ινδιγενών πληθυσμών σε επιχειρήσεις από κυβερνητικούς παράγοντες. Οι Ινδιγενείς πολλές φορές εκτοπίζονται από, τις, από τους αγρούς τους για τον λόγο αυτό αυτό είναι ένα πρόβλημα το οποίο θα στο οποίο θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή. Η βιομηχανία φινικελαίου σχετίζεται επίσης με έντονες παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων μεταξύ των οποίων και η και η παιδική εργασία μεταξύ των 7 εκατομμυρίων εργαζομένων στον τομέα υπάρχουν και εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά. Τα παρά, παράνομα προϊόντα επίσης εισάγονται στην εφοδιαστική αλυσίδα δημιουργώντας τεράστια κέρδη για πολυεθνικές επιχειρήσεις, καταστρέφοντας παράλληλα τη ζωή ανθρώπων. Ε, γι' αυτό ευθύνεται η μη βιώσιμη παραγωγή φινικελαίου. Αυτό που έχει γίνει μέχρι στιγμή από τις πολυεθνικές σε εθελοντικό στο επίπεδο δεν αρκεί για να επιτευχθεί ο στόχος πρέπει να σταματήσουν να συνεργάζονται με προμηθευτές που δεν πληρούν κάποια πρότυπα. Πολλές φορές δεν έχουμε επαρκή αναθεώρηση, εξέταση της τήρησης κάποιων προτύπων. Χρειαζόμαστε συνεπή κριτήρια και την συνεπή τήρησή τους. Γι' αυτό ζητούμε και την τήρηση σαφών διαδικασιών χορήγησης πιστοποίησης. Με βάση κάποια εθελοντικά προγράμματα οι εταιρείε έχουμε μια επαρκή τεκμηρίωση του τι κάνουν οι εταιρείε όσον αφορά τα ορυκτά συγκρούσεων. Ζητούμε ένα ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο θα διασφαλίζει πως ολόκληρη η εφοδιαστική αλυσίδα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα συνεισφέρει στο φαινόμενο της αποψήλωσης. Επίσης θα σώμαστε υπέρ μιας επακόλουθης νομοθεσίας Τέλος, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στην requires Σημειώνστε και τα ε, αναγκαία συστήματα πιστοποίησης. Ως καταναλωτές έχουμε την ευκαιρία να εξετάσουμε και τα πολλούμενα προϊόντα σε διάφορα σούπερ μάρκετ, εξετάζοντα ποιο είναι το περιεχόμενο των προϊόντων αυτών με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Δηλαδή, κάθε παραγωγό μπορεί επίση να συμβάλλει στην μείωση τη κατανάλωση φινικέλου, εφόσον χρησιμοποιεί τα προϊόντα αυτά. Ευχαριστώ πολύ ο Πρόεδρο και θα ακολουθήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ο κ. Τίλστρα. επιτρέψτε μου να προτείνω να δώσετε το λόγο στον ε, συναδελφό μου και εγώ θα συμπληρώσω τα όσα ε, έχει να σας πει. Ευχαριστώ και καλημέρα σας. Δράσεις για το φινικέλαιο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή γνωρίζει και την διασύνδεση μεταξύ καλλιέργειας φινικελαίου και αποψήλωσης δασών. Υπάρχει ωστόσο η αρχή της μη διάκρισης, την οποία γνωρίζετε καλά. Το φινικέλαιο συνδέεται σε ορισμένα μέρη του κόσμου με την αποψήλωση, αλλού γίνεται αποψήλωση ε, λόγω άλλων προϊόντων. Τίθεται ερώτημα λοιπόν γιατί ε, βάζουμε στο στόχαστρο αυτό το προϊόν και όχι κάποια άλλα. Νομίζω ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να ληφθεί υπόψη. να είμαστε ξεκάθαροι και σε ό,τι αφορά τις διατυπώσεις, διότι βιώσιμο φινικέλαιο σημαίνει άλλα πράγματα για διαφόρους και άλλα για διαφόρους. Ε, κριτήριο πρέπει να είναι η πρώτερη χρήση της γης, διότι το φινικέλαιο καλλιεργείται σε περιοχές όπου πριν ήταν δάση. Αυτό δεν προκύπτει όμως αυτομάτως από τη χρήση του όρου ε, βιώσιμο ή με βιώσιμο τρόπο καλλιεργημένο φινικέλαιο. Πρέπει λοιπόν και αυτό να ληφθεί υπόψη στην σύνταξη της γνωμοδότησης. Για τα βιολογικά καύσιμα, εξετάστε την οδηγία ανανεώσιμων ενεργειών. Φινικέλαιο που χρησιμοποιείται για την παραγωγή βιολογικού ντίζελ οφείλει να σέβεται ορισμένα κριτήρια μεταξύ αυτών και να μην καλλιεργούνται τα φινικόδεντρα δηλαδή σε πρόσφατα αποψηλωμένες εκτάσεις. Να λάβετε υπόψη και τις διάφορες οικειοθελείς πρωτοβουλίες Consumer Goods Forum στο οποίο συμμετέχουν πολλές μεγάλες διεθνώς γνωστές μάρκες και έχουν αποφασίσει zero deforestation, μηδενική αποψήλωση και ένα εργαλείο που πρόσφατα ε, ενέκρινε ο ΩΣΑ για τις υπεύθυνε ε, εφοδιαστικές αλυσίδες γραφτικών προϊόντων. Σε ό,τι αφορά τις FTA, τι συμφωνίες δηλαδή, αυτές συμφωνίες με την Μαλαισία και ε, οι διαπραγματεύσεις που συνεχίζονται με την Ινδονησία ασφαλώς και έχουν ε, σημαντική βαρύτητα εδώ και θα βάλουμε και κεφάλαιο για το βιώσιμο εμπόριο στις συμφωνίες αυτές. Θα μιλήσουμε την Ινδονησία να δούμε σε ποιο βαθμό θέματα που έχουν σχέση με το φινικέλαιο αλλά και γενικότερα με την διατήρηση της βιοπικιλότητας και των εργασιακών δικαιωμάτων, κατά πόσο λοιπόν τέτοια θέματα θα πρέπει να ενταχθούν στη συμφωνία αυτή. Γνωρίζετε όμως ότι βρισκόμαστε σε πρώιμο στάδιο των διαπραγματεύσεων αυτών. Ευχαριστώ. Ο έτερος της Ευρωπαϊκής Επιτροπή. Αν μπορώ να συμπληρώσω κάτι. Πρώτα, για την αποψήλωση δασών. ορισμένη εξ ημών ορθώς αναφέρατε το έργο, το οποίο έχουμε κάνει τα τελευταία 10-12 χρόνια, Έχουμε κάνει μεγάλη προσπάθεια για να επισημένονται τα προϊόντα αυτά, προϊόντα και παράνομης, παράνομης ξύλευσης. Η παράνομη υλοτομία είναι πάντως ένα από τα θέματα που συζητούνται μέσα στην, στα ζητήματα της αποψήλωσης και η Στατική της Ένωσης και το 7ο πρόγραμμα δράσεων ζητούν από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να ε, θεσπίσει ένα ε, σχέδιο δράσης για την ε, αποψήλωση δασών. Πρόσφατα έχουμε αναθέσει μια ανεξάρτητη μελέτη για να δούμε την δυνατότητα να αυξήσουμε τις δράσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να αντιμετωπιστεί η αποψήλωση καθώς και η ε, επιδείνωση της κατάστασης των δασών. Και θα τα θέσουμε αυτά τα επόμενα χρόνια ως θέματα. Ιδίως τώρα για το φινικέλαιο, πολλοί από εσά αναφερθήκατε στα αρνητικά, στις αρνητικές πτυχές της παραγωγής του φινικελαίου. Από την άλλη μεριά είναι σωστό να πει κανείς ότι πρόκειται για μια μεγάλη βιομηχανία, επομένως συνδέονται με αυτήν πολλά οικονομικά συμφέροντα και αποτελεί βεβαίω και πηγή εισοδήματο για τις αφορόμενες χώρες. Ασφαλώς αναγνωρίζουμε απολύτως όλες τις περιβαλλοντικές δυσμενείς επιπτώσεις που επιφέρει η παραγωγή φινικελαίου. Αυτό που θα κάνουμε είναι να ξεκινήσουμε σύντομα μια ειδική μελέτη για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καλλιέργειας φινικελαίου. Αυτή θα περιλάβει μια σε βάθος ανάλυση των υφιστάμενων προτύπων βιωσιμότητας. Ορισμένοι από εσά άλλωστε αναφερθήκατε σε αυτά. Αυτά θα επανεξεταστούν στην μελέτη αυτή και αυτό θα μας βοηθήσει να εξετάσουμε τι μπορούμε ενδεχομένω να κάνουμε σχετικά με το φινικέλαιο και με το ευρύτερο θέμα της αποψήλωσης τους επόμενους μήνες και χρόνια. Δύο λοιπόν πληροφορίες που ήθελα να θέσω υπόψη σας. Thanks And Ευχαριστώ. Κύριε Σιγητά. Ή μάλλον συγγνώμη κύριε Σιγητή. Να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους για τη συνεισφορά τους. Νομίζω ότι βρισκόμαστε στη σωστή άγουσα. Επομένως, θα προχωρήσουμε τις εργασίες μας και ελπίζω ότι θα καταφέρουμε να έχουμε το συντομότερο δυνατόν μια γνωμοδότηση με την οποία θα συμφωνούν περισσότερο. περισσότεροι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ την έκθεσή σας. Θα συνεχίσουμε να τη συζητούμε στις 5 Δεκεμβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Οπότε κλείνω το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Περνάω στο 9 της ολοκληρωμένης πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική. Πρόκειται για μια γνωμοδότηση για την ΑΦΕΤ και την ΕΝΒΗ για μια έκθεση. για μια ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει πολλές συνέπειες επίσης για το εμπόριο γι' αυτό και θα προβούμε σε μια γνωμοδότηση οπότε δίνω κατευθείαν τον λόγο στον εισηγητή David Martin Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε όπως γνωρίζουν οι συνάδελφοι, οκτώ χώρες καλύπτονται από την Ακτική, συμπεριλαμβανομένων δύο κρατών μελών της, Ευρω... μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή τη Δανία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία, τη Δανία, με, με την έννοια της Γρυλανδίας που ανήκει στη Δανία. Ως γνωστό, η κλιματική αλλαγή απειλεί την άγρια πανίδα στην περιοχή, αλλά ταυτόχρονα δημιουργεί νέες ευκαιρίες για οικονομική δραστηριότητα και επενδύσεις. Το λιώσιμο των πάγων δημιουργεί νέες διαδρομές ταυσιπλοείας αλλά ευνοεί επίσης νέες τουριστικές δραστηριότητες. Αυτό εξηγεί την στρατηγική σημασία που απέκτησε η Αρκτική Βλέπουμε λοιπόν ότι διάφορες χώρες και από την Ασία, μεταξύ των οποίων η Κίνα, έχουν στείλει παρατηρητές στην... για την Αρκτική. Εδώ όμως θα μιλήσουμε μόνο για τα εμπορικά και τις εμπορικές πτυχές της, εμπο... της της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην Ακτική. Όλες οι εμπορικές δραστηριότητες θα πρέπει να γίνουν με βιώσιμο τρόπο, με πλήρη σεβασμό προς τις συνδυγενείς κοινότητες. Δεύτερον, σύμφωνα ελεύθερου εμπορίου θα πρέπει να διασπαλίζουν πως οι αρχικές χώρες πληρούν υψηλά περιβαλλοντικά πρότυπα, όρους βιώσιμης αλληλείας. Αυτό έχει παραδείγματο χάρη για την ΣΥΤΑ και τις σχέσεις συμφωνίες μεταξύ Νορβηγίας και Ισλανδίας όσον αφορά τη χρήση φυσικών πόρων. κατόπιν πίεσης του παρόντος κοινοβουλίου έχουμε τήρηση τέτοιων μέτρων παρόμοια υιοθετήθηκαν επίσης από τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Ρωσία για τη διατήρηση της άγριας πανίδας στην περιοχή και των οικοσυστημάτων. Σχεδιάζω να καταθέσω κάποιες τροπολογίες που δεν μπόρεσα να περιλάβω στην πρωτότυπη γνωμοδότηση. Θα ήθελα να ζητήσω uh, δεσμευτικά πρότυπα, ευρύτερη, ευρύτερα εργαλεία χρηματοδοτικής συνεργασίας και επίσης θα καταθέσω μια τροπολογία για πρότυπα μεταφοράς διαθαλάσσης με δεσμευτικές απαιτήσεις για πλοία που λειτουργούν, που ταξιδεύουν στην Αρκτική και στην Ανταρκτική. Επίση θα ζητηθεί από την Γρυλανδία να... Θα, ήθελα να ζητηθεί από την Γρήλανδία να εφαρμόσει μια βιώσιμη αλληλεία στα χωρικά της ύδατα. Το περιβαλλοντικό στοιχείο είναι επίσης ένα άλλο στοιχείο στην, ε, όσον αφορά την Αρκτική. Εγώ εστίασα σε αυτά που ανέφερα μέχρι στιγμής. Πιστεύω πως αυτό είναι σημαντικό επειδή και σωστό, αλλιώς θα είχαμε κάποιο πρόβλημα με κάποια άλλη επιτροπή, οπότε δίνω το λόγο στην, στον σκιώδη, στη σκιώδη μάλλον. Η σκιώδη Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον εισηγητή μας ε, συνάδελφο David Μάρτιν για το σχέδιο και τις προτάσεις του. Επιθυμώ να προσθέσω ορισμένα στοιχεία. Αρχίζοντας από το σχέδιο για μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή πολιτική για την Αρκτική. Εδώ σημασία έχει να πούμε ότι η επικείμενη Φιλανδική Προεδρία του Αρκτικού Συμβουλίου 2017 έως 2018, στην οποία αναφέρθηκε ήδη ο Ντέβιτ, προσφέρει σημαντική ευκαιρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να αναπτύξει μια αρκτική πολιτική. Επίσης, ενώ η 16η διάσκεψη κορυφής που έγινε στις 13 Δεκάτου το λίγων ημερών δηλαδή, ο Καναδά και η Ευρωπαϊκή Ένωση συμφώνησαν να συνεργαστούν στενά με το Αρκτικό Συμβούλιο και νομίζω ότι θα πρέπει να αναμένουμε να λάβει την πλήρη απόφασή του το Αρκτικό Συμβούλιο για να δεχθεί την Ευρωπαϊκή Ένωση ως πλήρη παρατηρητή και αυτό θα γίνει στην κοινή διακήρυξη. Και σε ό,τι αφορά τη γνωμοδότηση της ΙΝΤΑ, της Επιτροπής μας δηλαδή, για την έκθεση, νομίζω ότι πρέπει να τονίσουμε την σημασία της εμπορικής πολιτικής της Ένωσης ως εργαλείο για να προωθηθούν ε, σημαντικές δεσμεύσεις και στόχοι για το περιβάλλον. Και ε, το ίδιο όπως οι ορισμένες FTA που έχουν ε, συναυθεί τελευταία, μεταξύ αυτών και η ΣΕΤΑ. Σημαντική, σημαντικό είναι επίσης το θέμα του ανοίγματο νέων οδών ναυσιπλοείας. Θα πρέπει εδώ να είμαστε ικανοποιημένοι από τα κεφάλαια της ΣΕΤΑ για το διεθνές εμπόριο και τις δημόσιες προμήθειες. Εγώ βεβαίως θα καταθέσω τροπολογία σχετικά με την έννοια ότι η συμμετοχή των ευρωπαϊκών εταιριών στην ε, καναδική αγορά δημοσίων προμηθειών θα έχει θετικές επιπτώσεις και ε, στην ε, ευρωπαϊκή ναυπική βιομηχανία και αυτούς που φτιάχνουν παγοθραυστικά σκάφη. Δεν θυμόμαι τον αριθμό της παραγράφου, αλλά αυτό που προτείνω είναι να τονίσουμε ότι Καναδάς και Ευρωπαϊκή Ένωση επανεπιβεβαίωσαν την δέσμευσή τους ενίσχυση της συνεργασίας τους στην Αρκτική. Και στην κοινή διακήρυξη της 16ης ε, ε, διάσκεψης κορυφής θα πρέπει να, να, να, μνημονευτεί και αυτή. Τέλος, στην παράγραφο όπου μιλούμε, πρόκειται την παράγραφο 5, μπορούμε να πούμε ότι θεωρούμε ότι η συμπερίληψη των διατάξεων αυτών θα πρέπει να είναι αναπόσπαστο μέρος οποιασδήποτε μελλοντική FTA, δηλαδή σε βάθος ε, εμπορικής συμφωνίας, που θα συνάψει η Ευρωπαϊκή Ένωση με τους ε, αρκτικούς εταίρους της. Εν ευθέτω χρόνο θα καταθέσω τις τροπολογίες αυτές και πάντως σας ευχαριστώ, David, για το σχέδιο. Ευχαριστώ, λέει ο Πρόεδρος, και Τώρα εξ ονόματος της ομάδας ECR. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ο κύριος Ζαχραντήλ. Ξέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει συνεισφέρει σημαντικά ως παράγον στην περιοχή της Αρκτικής και όσον αφορά τη δέσμευσή της ως προς την περιοχή και ως προς την πολιτική σε πολλοί τομεί στην αλληλεία, στους φυσικούς πόρους, ε, στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην έρευνα. Συνεπώς, αυτή η γνωμοδότηση είναι σαφέστατα απαραίτητη. Να επισημάνω κάποια σημεία. Πρώτον, νομίζω συμφωνώ με τον εισηγητή που τονίζει ότι υπάρχουν ευκαιρίες για οικονομική ανάπτυξη της περιοχής και ε, προπτικές επενδύσεων μέσω κατάλληλης εκμετάλλευσης των ενεργειακών πόρων, πετρελαίου και φυσικού αερίου. Ένα μόνο ίσως θα πρέπει να προσθέσουμε. Σίγουρα δεν θα είναι εύκολο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας το γεγονός ότι υπάρχουν περιορισμένες υποδομές, υπάρχουν περιορισμοί ανάλογα με την κάθε εποχή, λόγω του πάγου ε, και φυσικά ε, η περιοχή είναι παγωμένη και κατά την θερινή περίοδο. Στο σημείο 7 ο εισηγητή αναφέρεται Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου μεταξύ Ισλανδίας και Κίνας. Και αυτό είναι κάτι το οποίο σαφώς και πρέπει τρόπο την να μας απασχολήσει. Γνωρίζουμε ότι υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για, της Κίνας για την περιοχή και η συμφωνία μεταξύ Ισλανδίας και Κίνας μπορεί να αποτελεί ε, το πρώτο βήμα που κάνει το Πεκίνο προκειμένου να έχει καλύτερη πρόσβαση σε γραμμές ναυσιπλοείας μέσω της Αρκτικής και της εκμετάλλευσης των φυσικών της πόρων. Θα πρέπει λοιπόν να παρακολουθούμε και τις εξελίξεις εκεί. Και τρίτον, η Ρωσία. Μία ακόμα σημαντική δύναμη που έχει και το 50% περίπου της Αρκτικής. Οι σχέσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης Ρωσίας νομίζω είναι γνωστές αυτή τη στιγμή. Είναι σχεδόν ψυχρές. Δεν υπάρχει εμπορική συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας. Επομένως, οι δυνατότητες που έχουμε να παρακολουθήσουμε και να επηρεάσουμε τις δραστηριότητες του στην περιοχή είναι μάλλον περιορισμένες. Βεβαίως, η Αρκτική είναι μία από τις τελευταίες διεθνείς περιοχές στις οποίες υπάρχει τουλάχιστον τομεακός διάλογος μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ρωσίας και θα πρέπει να το εκμεταλλευτούμε αυτό για να παρακολουθούμε και πάλι τις εξελίξεις και να χρησιμοποιήσουμε και αυτή τουλάχιστον την πλευρά για να μπορέσουμε να επηρεάσουμε σε όποιο βαθμό μπορούμε τα ρωσικά συμφέροντα και δραστηριότητες στην περιοχή. Αυτά προς το παρόν. Συγχαρητήρια για το σχέδιο γνωμοδότηση. Προσβλέπω στη συνεργασία με το συντάκτη της γνωμοδότηση ώστε να την ολοκληρώσουμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο Χέλμουντ Σόλτ. Ευχαριστώ πολύ, Μπέντ. Ευχαριστώ με τη σειρά μου τον εισηγητή. Είναι σημαντική η γνωμοδότηση που έχει συντάξει. έχω κάποια σχόλια και ως ε, πολιτική ομάδα θα καταθέσουμε και τροπολογίες. Ας έχουμε υπόψη ότι το Μάρτιο του 2016 επιτύχαμε νέο αρνητικό ρεκόρ σε ό,τι αφορά το μέγεθος του πέρμαφρος, του, της κάλυψης από πάγους δηλαδή της Αρκτικής, αρνητικό ρεκόρ. Ό,τι έχουμε συζητήσει λοιπόν για εμπορικά και τέτοια Ωστόσο, κυριαρχεί το ζήτημα του περιβάλλοντος. Ευχαριστώ τη Γενική Διεύθυνση Ερευνών ή Μελετών του Ευρωκοινοβουλίου που έχουν εξυπηρετήσει και την Επιτροπή Εξωτερικών και άλλες κοινοβουλευτικές επιτροπές, δηλαδή ε, δημοσιεύοντας μια μελέτη για την Αρκτική και στη σελίδα 29 της μελέτης αυτής αναφέρονται οι προτεραιότητες των εθνικών στρατηγικών για την Αρκτική. Ως παράδειγμα, μόνο τρεις. Μιας και μιλούμε για εμπορικά θέματα. Πρώτον, Δανία, Φερόες και Γρυλανδία. Σημαντικές για την αποκατάσταση του περιβάλλοντος και του κλίματος. Σουηδία, Προστασία περιβάλλοντος, πρώτη προτεραιότητα και για την οικονομική ανάπτυξη και διεθνή συνεργασία. Ακόμα και οι Ηνωμένε Πολιτείε λένε ότι χρειάζεται προστασία του ακτικού περιβάλλοντος και των φυσικών του πόρων. Τα λέω αυτά για να καταστήσω σαφές ότι όλοι τάσσονται υπέρ της ανάγκης προστασίας του περιβάλλοντος, της βιωσιμότητας ή της αηφορίας της ε, περιοχής της Αρκτικής. Γι' αυτό και εμείς ως ενωτική αριστερά θέλουμε να μπει μια τέτοια διάσταση στην ευρωπαϊκή πολιτική για θέματα αρκτικής, την διατήρηση δηλαδή της αρκτικής ως αυτού που είναι, δηλαδή ένα μοναδικό φυσικό περιβάλλον και όχι ένα περιβάλλον μες στο οποίο μπορεί να συνεχίσετε η επιχειρηματική δραστηριότητα απρόσκοπτη. Χρειαζόμαστε λοιπόν πιο φιλόδοξα έργα, πιο φιλόδοξα σχέδια από αυτά που ακούμε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και από την ΥΠΑΤΗ εκπρόσωπο και αντιπρόεδρο της Κομισιόν. Νομίζω συμφωνούμε ότι αν συμβεί για παράδειγμα μια πετρελοκυλίδα στην Αρκτική θα είναι οι συνέπειες απρόβλεπτες και αδύνατον να αποκατασταθούν. Γι' αυτό θα πρέπει να πάρουμε το παράδειγμα της Ανταρκτικής, όπου έχει θεσπιστεί μεγαλύτερη περιοχή προστασίας του θαλάσσιου περιβάλλοντος. Συμφωνήθηκε μάλιστα πριν από λίγες εβδομάδες. Και αυτό θα πρέπει να οδηγήσει και μας να παγώσουμε όλες τις επιχειρηματικές δραστηριότητες που έχουν σχέση με εξόρυξη ορυκτών, πετρελαίου σε θαλάσσιες περιοχές της Αρκτικής ή κάτω από το έδαφος της Αρκτικής όπου χρησιμοποιείται και αργό πετρέλαιο για τα πλοία τα οποία διέρχονται από εκεί το ίδιο πρέπει να προστατεύσουμε και την, τα αλλιεύματα, δηλαδή να πάυσει η αλληλευτική δραστηριότητα στα ύδατα της Αρκτικής. Χρειάζεται δηλαδή να απαγορευτεί απολύτως η αλληλευτική για να μπορέσουν να ανακάμψουν τα αλλιεύματα και να απαγορευτεί η διέλευση δεξαμενοπλοίων. Πρέπει να ενισχυθεί και η ε, διάσταση αυτή στις πολιτικές των ε, χωρών που συνορεύουν με την Αρκτική και να μην προωθούνται οι επιχειρηματικές δραστηριότητες εξόριξης ρηκτών κλπ. και να βελτιωθεί η συνεργασία μετά την χωρών της Αρκτικής. Ευχαριστώ. Εσείς κύριε Τάκουλα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι έχουμε και κάποια παιδιά εδώ από τη Φιλανδία. Υπάρχει ε, και φιλανδική καμπίνα. Θα πω δύο λόγια στα φιλανδικά λοιπόν. Εγώ είμαι από την Αρκτική. Εντάξει, όχι ακριβώς, από τη Λαπωνία, στη Φιλανδία. Δίπλα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει πολιτική για την Αρκτική. Χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε πολλές προκλήσεις και η περιοχή της Αρκτικής ε, θα αντιμετωπίσει και πολλές προκλήσεις στο μέλλον. Επομένως πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερως. Ένας τρόπος λοιπόν να το κάνουμε αυτό είναι να δούμε και τι γίνεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Φιλανδία, η Δανία και η Σουηδία είναι οι χώρες οι οποίες συμμετέχουν άμεσα ε, στην περιοχή της Αρκτικής. Είναι χώρες της Αρκτικής γιατί έχουν αυτή τη σχέση, τη γεωγραφική. Επομένως πρέπει να λάβουμε υπόψη και τη βόρεια διάσταση στην Αρκτική περιοχή. Είναι επίσης πάρα πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη και ε, το γεγονός ότι είναι ευάλωτη η φύση στην περιοχή ε, είναι πολύ ευάλωτο το περιβάλλον και αυτό το επεσήμανε και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην πρότασή της. Ε, έχει αναφερθεί στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής και το γεγονός ότι το περιβάλλον είναι πάρα πολύ ευάλωτο εκεί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν να υπάρχει βιώσιμη υποδομή ε, στην Αρκτική και να γίνει με βιώσιμο τρόπο, ώστε να έχουμε ανάπτυξη ε, και να έχουμε επενδύσεις με βιώσιμο τρόπο. Πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψη και τη συμμετοχή της Ρωσίας στη συνεργασία. Οι κυρώσει ε, της Ρωσίας έχουν κάπως παραγωνίσει τη Ρωσία, αλλά δεν θα πρέπει να ε, λησμονούμε ότι όλοι πρέπει να δεσμευθούμε για την περιοχή και να υπάρχει εταιρική σχέση με τη Ρωσία. Η Αρκτική είναι μια περιοχή που έχει γεωπολιτική σημασία για την ε, Ρωσία, επομένως πρέπει να υπάρχει καλή συνεργασία, διότι μπορεί να είναι αμοιβαία επωφελής. Συνεπώς, κύριε Πρόεδρε, ο φίλος μας ο Ντέιβιτ Μάρτιν είναι συγητής. Γνωρίζω ότι είναι εξοικειωμένος με την περιοχή και ε, τον ενδιαφέρει να υπάρχει μια ισορροπημένη γνωμοδότηση για αυτή την όμορφη αλλά πολύ ευάλωτη περιοχή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την περιοχή της Αρκτικής, ώστε να την φροντίσουμε και να μπορέσουμε ε, να την εκμεταλλευτούμε ε, σωστά. Χρειαζόμαστε λοιπόν βιώσιμες λύσεις βιώσιμες οικονομικές λύσεις και όπως ε, ανέφερα επανειλημμένως και κατάλληλες υποδομές στις οποίες θα μπορέσουμε να τις βασίσουμε. Κάποιες σκέψεις λοιπόν και να πω ότι ευχαριστώ πολύ για τη γνωμοδότηση. Αυτά ευχαριστώ. Ευχαριστώ και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης στον κύριο Πίτερσεν. Λειτουργεί. Ναι. Ευχαριστώ. Είμαι σύμβουλο σε θέματα της Αρκτικής στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερική δράση και ευχαριστώ που μου δίνετε το λόγο. Υπάρχει μια κοινή δήλωση η οποία δημοσιεύτηκε τον Απρίλιο, η οποία στόχο έχει να εξισορροπήσει ακριβώς όλα όσα αναφέρατε κι εσείς και οι ομιλητές εδώ στην Επιτροπή, αλλά και σε άλλε επιτροπέ ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η κλιματική αλλαγή πιέζει ιδιαίτερα. Γίνονται λοιπόν προσπάθειες ώστε να υπάρχει και πρόληψη αλλά και προσαρμογή και να μετριάσουμε τα αποτελέσματα. Θέλουμε να προστατεύσουμε το περιβάλλον αλλά ε, σαφώς ε, λαμβάνουμε υπόψη και το σχόλιο που έκανε ο τελευταίος ομιλητής ε, εδώ Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην περιοχή, είναι μια ε, περιοχή με μεγάλη ποικιλομορφία, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που ζουν στην περιοχή και μας ζητούν να ε, την προφυλάξουμε. Επομένως, ε, θεωρώ ότι υπάρχουν μεγάλη διαφορά μεταξύ της Αρκτικής, στην οποία ζουν, και της Ανταρκτικής, στην οποία ζουν ελάχιστοι άνθρωποι. Είναι, λοιπόν, μια διαδικασία στην οποία πρέπει και να προστατεύσουμε και να προλάβουμε αρνητικές συνέπειες και να υπάρχει ταυτόχρονα και βιώσιμη ανάπτυξη της περιοχής. Η συνολική μας αίσθηση σε σχέση με τις προτάσεις που γίνονται στη γνωμοδότηση είναι ότι ε, σίγουρα είναι χρήσιμες, από ό,τι αντιλαμβάνομαι υπάρχουν και κάποιες τροπολογίες τις οποίες ε, ε, θα καταθέσει και ο ίδιο ο εισηγητή. αλλά θα πρέπει να γνωρίζετε ότι και εμεί παρακολουθούμε τις εργασίες. Ε, υπάρχει η Επιτροπή Αλληλείας, η Επιτροπή περιφερειακή ανάπτυξη και φυσικά και η Επιτροπή Περιβάλλοντος που παρακολουθούν το ζήτημα. Θα ήθελα επί, την ευκαιρία, επί τη ευκαιρία να επιστήσω την προσοχή σα και σε κάποιε συγκεκριμένε πτυχέ. Υπάρχουν εταίροι στην Αρκτική, το λέτε και εσεί στη γνωμοδότησή σα. Ε, τους οποίους δεν μπορούμε να επηρεάσουμε και τόσο και κάποιους άλλους που μπορούμε να επηρεάσουμε. Επομένως, πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ τι σήματα θα αποστείλουμε ιδίω ε, ενώπιση και τη συνολική κατάσταση. Όπω είπαμε όμω και στην ανακοίνωση, ε, Έχουμε επαφές ε, με όλες τις χώρες της Αρκτικής, χώρες που δεν είναι της Αρκτικής αλλά έχουν συμφέροντα στην περιοχή, με την ευρύτερη περιοχή, με τους κατοίκους, με την κοινωνία των πολιτών, με τις επιχειρήσεις και ελπίζουμε ότι ε, θα φτάσουμε ε, στις λεπτομέρειες μιας ισορροπημένης προσέγγισης. Να σας ευχαριστήσω παρεπιπτόντος για το πολύ ενδιαφέρον έργο σας. Σίγουρα θα συνεισφέρει στη δουλειά μας. Μία ερώτηση, Χέλμουτ, παρακαλώ. Έχω μία ερώτηση προς την Επιτροπή. Προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αν κατάλαβα σωστά, πιστεύω πως δεν θα πρέπει να έχουμε μία προσεκτική προσέγγιση, αλλά μία γενναία προσέγγιση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις αυτές πρέπει να δράσουμε. Επειδή δεν μας απομένει χρόνος. Και όλη την ώρα μιλούμε για το ότι πρέπει να κάνουμε το ένα ή το άλλο. Πιστεύω πως είναι πρόταγμα η προσέγγιση μας στην περιοχή αυτή. Και πιστεύω πως αυτό πρέπει να είναι επίσης το μήνυμα του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής μας. Χρειαζόμαστε περισσότερο θάρρος. Θέλει η υπηρεσία εξωτερική δράση να απαντήσει. Είστε πολύ προσεκτικοί, περισσότερο προσεκτικοί από γενναίοι πιστεύω από πολλές απόψεις θα αντιμετωπίσουμε ακριβώς το ερώτημα αυτό. Γνωρίζω πως το κοινοβούλιο αυτό ήδη από το 2008 εξέφρασε μια γνωμοδότηση για μια συνθήκη για την Αρκτική χωρίς να λάβει πολύ προσοχή. Εμείς προσπαθούμε με τη γνωμοδότηση αυτή να στείλουμε το μήνυμα πως είμαστε έτοιμοι να δραστηριοποιηθούμε με διάφορους επικοδομητικούς τρόπους, αλλά αυτή η κοινή ανακοίνωση δεν θα διορθώσει το πρόβλημα της Αρκτικής από μόνη της. Δεν είναι η νομοθεσία που θα κάνει τη διαφορά, αλλά η δραστηριοποίηση των ανθρώπων που ζουν εκεί και η διάδραση που έχουμε με τα κράτη και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη. Το πνεύμα της κοινή ανακοίνωσης είναι να προσπαθήσουμε να επιτύχουμε μια ισορροπία, αλλά αυτή η ανακοίνωση για την Αρκτική δεν είναι ένας κατάλογος νομοθετικών μέτρων, αλλά ένας πολιτικός παλμός. και πιστεύω πως προσπαθούμε να επιτύχουμε την ισορροπία όσο το δυνατόν πιο επικοδομητικά μπορούμε. Και η απόκριση από την Αρκτική ήταν αρκετά θετική μέχρι στιγμή. Η δέσμευση της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο Συμβούλιο της Αρκτικής κατά τη συνεργασία με τα κράτη και τις περιφέρειες όπως θα ξέρετε σε όλη την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Υπάρχουν γενικέ διευθύνσει που εμπλέκονται στι διαπραγματεύσει για το κλίμα που λαμβάνουν χώρα τώρα στο Μάρακε. που προώθησαν αλλαγές στο πρωτόκολλο του Μόντρεαλ, που εγκρίθηκε στο Κιγκάλι πρόσφατα. Δηλαδή υπάρχουν διάφορε πρωτοβουλίες που βρίσκονται σαφώς στο πνεύμα αυτή της κοινή ανακοίνωση. Αφετέρου πρέπει να καταλάβουμε πως υπάρχει μια οικονομική εξέλιξη καθώς η περιοχή βρίσκεται υπό τον έλεγχο των αρκτικών κρατών. Εάν θέλουμε να την επηρεάσουμε, πρέπει να συνεργαστούμε μαζί τους. Νομίζω αυτό είπε και ο, ο Φιλανδό ομιλητής πριν. Εάν θέλουμε να ασκήσουμε επιρροή, δεν μπορούμε απλά να κλειστούμε, να απομονωθούμε σε γραφεία. Πρόκειται για μια ευαίσθητη ισορροπία και εκτιμώ πολύ αυτό που είπε ο κύριος Σούλτς φυσικά και προσμένουμε το πλήρες ψήφισμα του Κοινοβουλίου αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Και τώρα ο εισηγητής David Μάρτιν. Επ' αυτού νομίζω ότι προσεγγίζω την στάση της υπηρεσίας εξωτερικών δράσεων. Χρειάζεται πράγματι μια σε βάθος προσέγγιση. Είναι κάτι τόσο έφραυστο η Αρκτική. Πρέπει όμως να είμαστε και Να πούμε πρώτα ότι τα προβλήματα αλλαγής κλίματος που αντιμετωπίζει η Αρκτική δεν είναι το φταίξιμο της Αρκτικής, είναι τα θύματα η Αρκτική και ο κόσμος που ζει σε αυτήν. Δεύτερον, πρόκειται για έφραστα οικοσυστήματα που πρέπει να κάνουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τα προστατεύσουμε και να τα διατηρήσουμε, όπως είπε και ο Χάνου Τάκολα, αλλά και οι άνθρωποι των εξωτερικών δράσεων. Υπάρχουν άνθρωποι που κατοικούν, που ζουν εκεί και θέλουν να συναποτελούν μέρος του, του κόσμου. Τέλος, η επιρροή μας είναι περιορισμένη. Μόλις πρόσφατα ε, λάβαμε το καθεστώς του παρατηρητή στο Αρκτικό Συμβούλιο, η Ρωσία είναι μέγας παίκτης εκεί, ο Καναδάς είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος, η δική μας επιρροή είναι περιορισμένη. Πρέπει λοιπόν να στοχεύσουμε σε αυτά που μπορούμε πράγματι να κάνουμε. Έγιναν χρήσιμες προτάσεις όπως η κυρία Αντρικάιτεν, να χρησιμοποιήσουμε την ευκαιρία δηλαδή της Φιλανδικής Προεδρίας, πολύ χρήσιμο αυτό, να κάνουμε ό,τι μπορούμε και μέσω της συνεργασίας στην βάση της Συμφωνίας ΣΕΤΑ με τον Καναδά για να προωθήσουμε προοδευτικές πολιτικές και ιδίω σε διεθνείς οργανισμούς, πάλι όπως είπε η κυρία Αντρικίενε, την ε, διεθνή, ε, τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό και όλους τους άλλους ε, να επιβάλλουν δηλαδή υψηλά πρότυπα ασφαλείας για τις θαλάσσιες οδούς και να προσπαθήσουμε με κάθε τρόπο να προστατεύσουμε την Αρκτική. Από τις λίγες επαφές που έχω και εδώ έχουμε σε αντίθεση με την υπηρεσία εξωτερικών δράσεων, από τις λίγες επαφές που έχω με, για, με τους Ρώσους, αλλά έχω μιλώντας και με Φιλανδούς και άλλους, οι Φιλανδοί μου λένε ότι η Ρωσία συνεργάζεται πλήρως στο Αρκτικό Συμβούλιο και ότι η συνεργασία μαζί της είναι καλή μέσα στα πλαίσια αυτού του οργανισμού θα πρέπει να συνεχίσουμε ανεξαρτήτως του τι συμβαίνει σε άλλους τομείς. Βεβαίως, πόσες προσπάθειες χρειάζονται. Πρόκειται για έφθαστο οικοσύστημα που πρέπει να το προστατεύσουμε με ένα ε, τρόπο ε, που να είναι αποτελεσματικός, αλλά βεβαίως η επιρροή μας, όπως είπα, είναι περιορισμένη. Δεν είναι ε, όσοι θα θέλαμε να είναι. Ευχαριστώ πολύ, λέει ο πρόεδρος Μπέρντ Λάγκε. Το ψήφισμα του 2008, εξάλλου, δεν ήταν απόλυτα σαφές ότι ζητούμε συνθήκη. Προβληματιζόμασταν τότε επί της δυνατότητας να υπάρξει τέτοια συνθήκη. Παρ' όλα αυτά θα συνεχίσουμε το εγχείρημα. Τροπολογίες μπορούν να κατατεθούν έως τις 14 ενδεκάτου που είναι η ερχομένη Δευτέρα μέχρι τις 12 το μεσημέρι ακριβώς που θα είναι ψηλά ο ήλιος στις 5 Δεκεμβρίου θα επανέλθουμε εδώ στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ πολύ και τώρα έρχομαι στο υπαριθμό 10 την παρουσίαση μελέτης για την ευρωπαϊκή πολιτική, εμπορική συγγνώμη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το εμπόριο αγρίων ειδών. Η ε, κυρία Ντάφη είναι παρούσα και είναι καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο του Σέφιλντ και το σχέδιο μελέτης βρίσκεται και στην ιστοσελίδα της ίντα. Καλώς ήρθατε κυρία καθηγήτρια. Θα θυμάστε ότι είχαμε ένα εργαστήριο για το θέμα αυτό προ λίγων εβδομάδων και θα συνεχίσουμε την δουλειά αυτή με έκθεση της ε, κυρίας Μακλάκλιν Τώρα όμως θα εγκύψουμε στη μελέτη σας και θα σας δώσουμε 10 λεπτά για να την παρουσιάσετε. Ευχαριστώ πολύ και σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Έχω κάποιες διαφάνειες, ε, θα τις διατρέξω. Και εδώ έχουμε τη νόμιμη και την παράνομη διάσταση του εμπορίου αγριονιδών. Από ό,τι βλέπετε η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει πολύ σημαντικό ε, ποσοστό και ε, νόμιμων και παράνομων προϊόντων τα οποία εμπορεύονται εντό Ευρωπαϊκής Ένωσης. 641 εκατομμύρια ευρώ το 2014, αυτά είναι τα πιο πρόσφατα στοιχεία ε, και τα έχει συγκεντρώσει η τράφικ και έχουμε και εξαγωγές χαβιαριού, οι οποίες είναι πάρα πολύ σημαντικές. Επίσης βλέπουμε ότι η κατανομή των προϊόντων ε, τα οποία την χάνουν εμπορία και νομίμως και παρανόμως στην Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι κατά κύριο λόγο φάρμακα ε, από φυτικά προϊόντα, αλλά έχουμε και θηλαστικά, ερπετά, είναι πολύ μεγάλα τα ποσοστά, κυρίως για κατοικίδια, ασπόνδυλα κλπ η αξιολόγηση αυτού του εμπορίου είναι λίγο προβληματική. Δεν μπορούμε να κάνουμε διαχωρισμού μεταξύ νόμιμου και παράνομου εμπορίου και κυρίως των ειδών, διότι είναι πολλές φορές ε, το ένα μέσα στο άλλο και επομένως μπορεί να αλλάξει και πάρα πολύ ε, ο συσχετισμός και πολύ γρήγορα. Βάσει των στοιχείων όμως που μας δίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και η ανταλλαγή ε, πληροφοριών για το εμπόριο σε αγρία ε, έχουμε εδώ στη διαφάνεια, όπως βλέπετε, τις βασικές ε, διόδους από τις οποίες γίνεται το εμπόριο και τι γίνεται με τις εξαγωγές. Έχουμε νόμιμα και παράνομο εμπόριο, κυρίως ε, από και προς την Ασία. Έχουμε τέσσερις βασικές οδούς, από την Αφρική σε βασικούς κόμβους στην Ευρώπη. Έχουμε παράκτιο ελαφρεμπόριο στην Νότια Ευρώπη κυρίως, υπάρχει νοτιοανατολικό εμπόριο και υπάρχουν και χερσαίες οδοί. Ο βασικός μοχλών της αύξησης ε, και στο νόμιμο και στο παράνομο εμπόριο ε, τα τελευταία χρόνια είναι ότι οι άνθρωποι στις πιο εύρωστες ε, περιοχές, όχι απαραίτητα χώρες, αλλά σε πιο εύρωστες κοινότητες, έχουν συνηθίσει έναν τρόπο ζωής που έχει μεγάλη ζήτηση και για τρόφιμα και για δερμάτινα είδη και για φάρμακα ε, και έχουμε για παράδειγμα δέρμα ερπετών ε, για τη βιομηχανία της μόδας, αλλά επίσης και ζήτηση για προϊόντα άγριων ζώων, ε, για παραδοσιακά κινέζικα φάρμακα. Παραδείγματο χάρη για το χαβιάρι. Τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ενωμένο Βασίλειο, εισάγουν περισσότερο από όλους χαβιάρι αναφέρονται ε, στις άδειες του site της. Το site της έχει ζητήσει ένα παγκόσμιο σύστημα επισήμανσης. Το χαβιάρι είναι ένα από τα σπάνια παραδείγματος ε, ε μίας ε, ε, πρώτερης εγγραφής στους καταλόγους του site Τα περισσότερα βρίσκονται στο παράρτημα 1, το οποίο παράρτημα σημαίνει ότι υπάρχει πλήρης απαγόρευση εμπορίου, ενώ τα είδη που βρίσκονται στο παράρτημα 2 επιτρέπει νόμιμο έλεγχο και... Ε, είδη ε, τα οποία παρακολουθούνται ε, συστηματικά. Έχουμε λοιπόν ε, διαχειριστικές αρχές του site που παρακολουθούν διαχειριστικές αρχές τις οποίες έχει εγκρίνει ο site για παρακολούθηση. Μπορεί να υπάρχει επισήμανση ότι μπορεί το χαβιάριο ξύριγχου να θεωρείται ότι είναι νόμιμο και από ενώ πολλές φορές είναι παράνομο ο χαβιάρι. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε και κάποια κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, που θα ήταν εύκολο βέβαια να πούμε ότι ε, είναι τμήμα του προβλήματος αλλά ε, όλες οι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα μπορούσαν να κάνουν κάτι για να βελτιώσουν την κατάσταση. Είναι εισαγωγέας, εξαγωγέας Ευρωπαϊκή Ένωση και περιοχή από την οποία περνούν τα προϊόντα για να μεταφερθούν αλλού. Ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία ε, και οι κάτω χώρες είναι από τις χώρες που χρησιμοποιούνται περισσότερο ε, για διέλευση αυτών των προϊόντων, αλλά δεν αποτελούν και πολύ σημαντικού δείκτες για τους όγκους του παράνομου εμπορίου. Τα στοιχεία που έχουμε μπορεί να μας δείχνουν ότι σε κάποιες χώρες μπορεί να επιβάλλονται καλύτερα τα μέτρα παρακολούθησης, αλλά δεν μας δείχνουν τι ακριβώς συμβαίνει. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρόσφατα προσχώρησε στο site της το 2015 και συμμετείχε και στην COP17 ε, για πρώτη φορά φέτος. Και οι 20 προτάσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, έγιναν αποδεκτές από το site της. Υπάρχει λοιπόν ένα καλό ιστορικό το οποίο μπορούμε να συνεχίσουμε και να το ε, εμβαθύνουμε περισσότερο. Όσον αφορά τα μέσα εμπορίου, διότι με ρωτήσετε κυρίω για το εμπόριο, μπορούμε να τα χρησιμοποιήσουμε για νόμιμο και βιώσιμο εμπόριο, αλλά και για να αντιμετωπίσουμε και το λαθρεμπόριο. Ε, δεν μπορεί να υπάρξει βεβαίω επιτυχία εάν χρησιμοποιούμε μόνο εμπορική πολιτική. Τα εμπορικά μέσα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό με ευρύτερα μέσα αντιμετώπιση του ε, ε, εμπορίου αυτού, ε, γιατί είναι πολύ μεγάλο το φάσμα των λόγων για τους οποίους γίνεται παράνομο εμπόριο. Πρέπει να μειώσουμε την ένδυα και την ανισότητα στις χώρες καταγωγής, να μειώσουμε τη ζήτηση στις χώρες κατανάλωσης, να αντιμετωπίσουμε τη διαφθορά, το οργανωμένο έγκλημα, την ελληπή εφαρμογή και τις ε, χαμηλές ποινές. Όσον αφορά το νόμιμο εμπόριο, είναι πολύ σημαντική πηγή εισοδήματος ε, και βιώσιμης ε, ε, βιώσιμων δυνατοτήτων στις πιο φτωχές κοινότητες του κόσμου. Για παράδειγμα, το πρόγραμμα δράσης κατά του λαθρεμπορίου των άγριων ζώων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε ότι πρέπει να υπάρχει ανάγκη να δεσμευτούμε με τις αγροτικές κοινότητες για να αντιμετωπίσουμε τα αίτια της παράνομης αυτής δραστηριότητας θα πρέπει να δούμε για παράδειγμα τι μπορούμε να κάνουμε μέσω και των προγραμμάτων, όπως για παράδειγμα το Aid for Trade. Οι παγκόσμιες Αλυσίδε διανομής είναι ένας τρόπος για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε τα ε, διάφορα εμπορικά μέσα, αλλά ορισμένες φορές ε, στους ε, χώρους διατήρησης των άγριων τζών και πανίδας και χλωρίδας λέγεται ότι Υπάρχει πρόβλημα λόγω των φτωχότερων κοινοτήτων. Θα πρέπει λοιπόν οι φτωχότερες κοινότητες παραγωγή να πρέπει να ε, έχουν τις μεγαλύτερες απολαβές ε, από το εμπόριο αυτό και αυτό φυσικά θα συνεισφέρει με τις προσεγγίσεις που έχουμε για τις παγκόσμιες αλυσίδες. Για παράδειγμα, στην Νοτιοανατολική Ασία για το δέρμα πίθωνα ο κυνηγό θα πάρει περίπου το 0,5% της αξίας ε, μιας τσάντας με δέρμα πίθωνα που θα πουληθεί στην Ευρώπη. Ε, γίνεται μεταποίηση και όταν το δέρμα ε, γίνεται πλέον καταναλωτικό αγαθό, εκεί έχουμε το μεγαλύτερο κέρδος. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν θα μπορούσε να προσφέρει υποστήριξη για να δημιουργήσουμε ικανότητες ώστε να βοηθήσουμε τις τοπικές κοινότητες για να αποκομίζουν περισσότερα ωφέλη από το εμπόριο αυτό. Ε, ε συμφωνίες ελευθέρου εμπορίου και συμφωνίες GSPC έχουμε συμφωνίες με την Νότια Κορέα και συμφώνησαν να εφαρμόσουν και τη Συμφωνία Ελευθέρου Εμπορίου με το Βιετνάμ και αυτή τη στιγμή είναι σε διαπραγματεύσει με την Ιαπωνία. Σήμερα, πέραν από τη συμφωνία με το Βιετνάμ, δεν υπάρχει κάποια συγκεκριμένη αναφορά στο εμπόριο σε άγρια είδη, είτε νόμιμο είτε παράνομο. Ε, το να υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, λοιπόν, ίσως είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας βοηθήσει να έχουμε κάποιες εξελίξει στο μέλλον. Το ίδιο ισχύει και για τις πρωτομησιακέ συμφωνίες GSP και GSPC, για να μπορέσουμε να έχουμε και εκεί κάποια μέτρα τα οποία σχετίζονται με τα άγρια δώα. Η TTIP θα μπορούσε να ακολουθήσει και το παράδειγμα της TPP για να μπορέσουμε να έχουμε συγκεκριμένα πράγματα για το λαθρεμπόριο των αγριών και να υπάρχει και διαφάνεια για να μπορέσουν οι εθνικές κυβερνήσεις να εφαρμόσουν νομοθεσία για να υποστηρίξει νόμιμο εμπόριο αγριών και να αντιμετωπίσει το παράνομο εμπόριο. Οι βασικές προκλήσεις παρά το γεγονό ότι η παγκοσμία ασφάλεια και η σχέση μεταξύ λαθρεμπορίου, οργανωμένου εγκλήματο ε, και τρομοκρατίας είναι αυτά τα οποία προσέχουμε περισσότερο αυτή τη στιγμή, κατά την άποψή μου υπάρχουν πιο πιεστικές ανάγκες και τομείς στου οποίου θα μπορούσε να επικεντρωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Παραδείγματο χάρη στον τομέα των μεταφορών η ανάγκη να έχουμε κάποιες συγκεκριμένες υποχρεώσεις και να μην υπάρχει λαθρεμπόριο αγρονιδών έχει αναγνωριστεί από τις παγκόσμιες μεταφερικές εταιρείες και πρέπει να υπάρχει συμμετοχή κυβερνητικών οργανώσεων. Υπάρχει μια δήλωση, μια, εθνική, μια διεθνής task force ε, έχει υπογράψει η COSCO, η Kenya Airways, η RATA, η ε, Διεθνής Οργάνωση ε, Μεταφορέων Κάργο, ε, και αυτό δείχνει ότι ο κλάδος αναγνωρίζει πάρα πολύ το πόσο σημαντικά είναι όλα αυτά και επίσης υπάρχουν και νέες, τροπολογίες στον τομέα, νέες πρωτοβουλίες συγγνώμη, στον τομέα των μεταφορών. Η USAID δεσμεύτηκε για πέντε χρόνια χρηματοδότησης για το πρόγραμμα Roots, ε, το οποίο έχει αναλάβει η μη κυβερνητική οργάνωση Traffic. Θα μπορούσαμε επίσης να ενισχύσουμε και τη συνεργασία στους τομείς αυτούς στον τομέα των μεταφορών. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό ε, στην Τελωνιακή Ένωση ή στο χώρο Σέγγεν. Και πάλι αυτό έχει σχέση με τη μεταφορά και την εφαρμογή της νομοθεσίας. Το περιβαλλοντικό έγκλημα πολλές φορές έχει διεθνή διάσταση. Το ηλεκτρονικό εμπόριο επίσης είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα μπορούσε να είναι ένας θετικός τρόπος να συνδέσουμε τους παραγωγούς και τους καταναλωτές. Αλλά επίσης ε, ε, πολύ συχνά χρησιμοποιείται και για λαθρεμπόριο αγριονιδών γιατί υπάρχει πολύ χαμηλός κίνδυνος να συλληφθούν ε, κυρίως μέσω της χρήσης ε, μέσων κοινωνικής δικτύωσης όπως το WeChat και το Alibaba. Η ανταλλαγή δεδομένων είναι πάρα πολύ σημαντική, αλλά αυτό που έχει περισσότερη σημασία είναι να χρησιμοποιήσουμε καλύτερα μηχανισμούς που έχουμε στη διάθεσή μας. Στη βάση δεδομένων EU Twix, για παράδειγμα, και όχι να αναπτύξουμε νέες βάσεις δεδομένων. Υπάρχουν μηχανισμοί και εργαλεία, αλλά πρέπει να χρησιμοποιούν αποτελεσματικά. Και τέλο, πρέπει να μειωθεί η ζήτηση. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει μια προσέγγιση που θα αποτενθεί στην κοινωνία. Χρειάζονται χρόνια για να υπάρξουν οποιαδήποτε αποτελέσματα, αλλά σίγουρα μπορεί να έχει αποτέλεσμα. Υπήρχε, για παράδειγμα, μείωση στη ζήτηση στο ελεφαντόδοντο το 1989 και στην Ευρώπη και στη Βόρεια Αμερική. Επομένω, οι εκστρατείε μπορούν να έχουν αποτελέσματα. Υπάρχουν κάποιε συστάσει στην έκθεση. Δεν ξέρω αν έχω χρόνο να σα τι αναφέρω. Αλλά η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να επικεντρωθεί στην εφαρμογή και ε, υλοποίηση των δεσμεύσεών τη. Θα πρέπει επίση να υπάρχουν πλατφόρμε ανταλλαγή δεδομένων που χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικό και οι μελλοντικέ ε, διαπραγματεύσει και παρούσε διαπραγματεύσει για συμφωνίε ελευθέρου εμπορίου μπορούν να περιλαμβάνουν διατάξει για το εμπόριο άγνων ειδών. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να υποστηρίξει επίση κατάρτιση για ε, οργανώσει παραγωγών, κοινωνικέ επιχειρήσει κλπ. για να υπάρχει μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία για τον, τα προϊόντα αυτά. Να υπάρχει το Aid Blending και το Aid for Trade. Είναι πολύ καλά μέσα τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν και όλα αυτά θα μπορούσαν να υποστηρίξουν την ανάπτυξη ηλεκτρονικού εμπορίου για να υποστηρίξουμε βιώσιμο νόμιμο εμπόριο και να συνεργαστούμε με οργανώσεις που μπορούν να βοηθήσουν για να αντιμετωπίσουμε το λαθρεμπόριο. Τέλος, η Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να αναπτύξει κατευθυντηρίες γραμμές για παράγοντες του ιδιωτικού κλάδου που συμμετέχουν ενεργά στο εμπόριο ειδών, να υπάρχουν έλεγχοι στα κέντρα αποστολής ε, και να μπορέσουν να είναι πιο νόμιμες οι μέθοδοι και επίσης να ε, μειώσουμε τη ζήτηση, διότι αυτές οι πρωτοβουλίες είναι οι πιο αποτελεσματικές για την αντιμετώπιση του λαθρεμπορίου αυτών των ειδών. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ κυρία καθηγήτρια για την ενδιαφέρουσα μελέτη. ο εισηγητής για την TTIP δεν είμαι πεπισμένος ότι θα έχουμε καν την ευκαιρία να διαπραγματευτούμε τέτοιου είδους κεφάλαιο για τη συμφωνία TTIP. Δεν είμαι διόλου βέβαιος ότι θα συνεχιστούν οι διαπραγματεύσεις. Παρ' όλα αυτά, στην, έκθεση, στην μελέτη σας μάλλον ε, περιλήφθηκαν σημαντικά και ενδιαφέροντα πράγματα. Και πρώτα ο David Μάρτιν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για την παρουσίαση. Δύσκολο να διαφωνήσει κανείς με τα συμπεράσματα που είναι πάρα πολύ λογικά. Έχω ίσως κάποια διευκρινιστικά. Το παράδειγμα του χαβιαριού είναι ένα παράδειγμα είδους όπου υπάρχει μια περιορισμένη απαγόρευση και όχι γενική απαγόρευση εμπορίου για την προστασία. Γιατί εκεί πρόκειται για προστασία και αγριών αλλά υπάρχει και εμπορική παραγωγή. Οι περιορισμένες απαγορεύσεις, αν κατάλαβα καλά, δεν αποδίδουν. Προτιμάτε πλήρης απαγορεύσεις. Ή μιλείτε για καλύτερη αποκάλυψη, detection δηλαδή, των ε, ε, ροών αυτών για τις Free Trade Agreements, συμφωνίες ελευθερών εμπορίου. Όλοι συμφωνούμε να μπουν, να, που μπαίνει κεφάλαιο για την προστασία της ε, άγριας ζωής στη συμφωνία με το Βιετνάμ. Ωστόσο παρόλα αυτά είμαι και κάπως επιφυλακτικός, δηλαδή τι διαφορά τελικώς θα επιφέρει στην πραγματικότητα. Αν εξετάσετε τα κεφάλαια ε, εμπορίου και ε, αεφόρου ανάπτυξη κλπ πολλοί ας πούμε ευρωβουλευτές δεν πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματικά αυτά και διερωτώ αν να περιλάβουμε και κεφάλαια για την ε, αδάμα στη ζωή, αν τελικώς θα αποδώσει τίποτε. Έχετε ίσως προτάσεις για να δούμε πώς θα μπορούσαμε ίσως να τα ενισχύσουμε τα κεφάλαια αυτά. Για τη συμφωνία με το Βιετνάμ, που είναι πράγματι μια θετική αφετηρία, αλλά θα χρειάζεται να συνεχιστεί στο μέλλον. Η καθηγήτρια, είναι πολύ ενδιαφέρουσε οι ερωτήσει σα. Προσωπικά, δεν τάσομαι υπέρ των πλήρων εμπορικών απαγορεύσεων. Μερικές απαγορεύσεις έχουν αποδώσει, αλλά όχι απολύτως. Και η σχεδόν αποκλειστική απαγόρευση του εμπορίου ε, ε, ελεφαντόδοντου έχει κάτι αποδώσει, αλλά δεν έχει σταματήσει τη λαθροθυρία. Η μείωση της ζήτησης είναι ο καλύτερος τρόπος. Βλέπε και την οργάνωση ΣΑΙΤΕΣ. Για την περίπτωση του χαβιαριού, νομίζω ότι η βελτιωμένη επιβολή, η βελτιωμένη επισήμανση, γιατί επιτρέπεται μικρή ποσότητα μόνο για προσωπική χρήση, που δεν χρειάζεται δηλαδή να είναι επισημασμένη ή να συνοδεύεται από έγγραφα σάιτες για το όνομα μου Χαβιάρη δηλαδή. Εδώ είναι καλύτερα να βελτιωθεί η επιβολή. Συμφωνώ επίσης ότι σε πολλές από τις συμφωνίες αντιλαμβάνομαι ότι αμφισβητείται η TTIP, αλλά και η FTA και οι συμφωνίες οικονομικής συνεργασίας περιλαμβάνουν και θέματα βιωσιμότητας όπως και η συμφωνία του Βιετνάμ και οι χώρες πρέπει να δείξουν, άλλωστε συμμετέχουν, υπογράφουν και μεγάλες ε, διεθνείς συμφωνίες. Νομίζω ότι είναι καλή η στόχη αυτή, πρέπει όμως να επιβάλλονται δεσμευτικά και να εγγράφονται και στις συμφωνίες, κάτι το οποίο διευκολύνει τις εθνικές κυβερνήσεις των χωρών που συμμετέχουν στις συμφωνίες αυτές να τα επιβάλλουν και στο εσωτερικό τα πράγματα αυτά και να εξηγήσουν γιατί. Άλλες ερωτήσεις? Όχι. Από τη δική μου πλευρά σχετικά με το κεφάλαιο για τις εμπορικές συμφωνίες. Το συζητήσαμε αρκετά σε βάθος ε, για τη συμφωνία με το Βιετνάμ και στη διάρκεια των διαπραγματεύσεων με την χώρα αυτή. Περιμένουμε τώρα την διέλευση της συμφωνίας από το Κοινοβούλιο. Μπορείτε να εξηγήσετε λίγο περισσότερο ποιες βρίσκεται ότι είναι οι ευκαιρίες που ανοίγει το κεφάλαιο αυτό ή τέλος πάντων οι δυνατότητες που προσφέρει. Διότι τώρα διαπραγματευόμαστε και με την Ινδονησία και με άλλες χώρες στην περιοχή αυτή του κόσμου. Και χρειαζόμαστε να έχουμε το απόλυτο πρότυπο για, τις, ε, για τέτοια κεφάλαια στις συμφωνίες αυτές. Δεύτερο, για τους συνοριακούς ελέγχους και την κατάσταση στα λιμάνια μας. Πού νομίζετε ότι σημειώνονται κάποια καλά παραδείγματα ή κάποια καλύτερα παραδείγματα αλλού και πώς μπορούν να βελτιωθούν οι συνοριακοί έλεγχοι. Όπως είπατε, χρειάζεται ένα απόλυτο πρότυπο, ένα gold standard. Όντω, η συμφωνία με το Βιετνάμ αποτελεί μια αρχή. Εκεί σημασία έχει η επιβολή. Στην περίπτωση του Βιετνάμ για το ICCWC. Κάποια ενίσχυση χρειάζεται ώστε να δημιουργηθεί η ικανότητα στη χώρα αυτή για να μπορεί να επιβάλλει τους ελέγχους αυτούς ως μια συνέχεια, ως ένα follow-up της εγγραφής των κριτηρίων αυτών και των κεφαλαίων αυτών στις συμφωνίες. Τώρα, σε ό,τι αφορά τους συνοριακούς ελέγχους, Εκεί αυτοί πρέπει να στοχεύσουν κυρίως την προστασία των εξωτερικών συνόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πρόσθετη έλεγχη βέβαια όταν το προϊόν εισέλθει ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι υπό τους, τους ε, κανόνες του ΠΟΕ επιτρέπονται οι εσωτερικοί έλεγχοι μετά την διέλευση δηλαδή από τα σύνορα, εφόσον υπάρχουν θέματα ε, διατήρησης περιβάλλοντος κλπ. Και μέσα στην ε, και μέσα στον χώρο Σέγγεν άλλωστε. Για παράδειγμα, κέντρα ε, κέντρα διανομής ταχυδρομικών δεμάτων κλπ. Εκεί ε, ίσως μπορεί η Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει νέους κανόνες για την επιθεώρηση των αποστολών στα ε, κέντρα αυτά. Ευχαριστώ, ο Πρόεδρος Ωραία, εδώ λίγη η συζήτηση του θέματος αυτού. Νομίζω ότι όλοι έχετε αντίγραφο του σχεδίου, το οποίο σχέδιο άλλωστε υπάρχει και στην ιστοσελίδα μας. Ευχαριστώ λοιπόν και πάλι, σας ευχαριστώ και εσάς κυρία Καθηγητή. Σε πέντε λεπτά αρχίζει η συνεδρία των συντονιστών, οι οποίοι βεβαίω είναι και κλεισμένων των θυρών. Και θυμηθείτε ότι αρχίζουμε μετά στις 2, δηλαδή νωρίτερα από ό,τι συνήθως. Ακριβώς λοιπόν στις 2 στην ε, παρούσα αίθουσα. Και σε 5 λεπτά αρχίζουν οι συντονιστές.